το μήνυμα του Προέδρου, ο οποίο δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα γιατί έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Αναλάβω λοιπόν εγώ την Προεδρία σήμερα το απόγευμα και προτείνω να ξεκινήσουμε στο, με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης που είναι ε, η έγκριση αυτή. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη ω έχει. Καμία αντίρρηση εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο έγκριση των πρακτικών της συνειδρύσης, τη συνεδρία της 21ης και 22ης Ιανουαρίου. Αν δεν υπάρχουν σχόλια ή αντιρρήσεις, προτείνω να εγκριθούν. Περνάμε και μετά από αυτό στο σημείο 3, που είναι οι ανακοινώσει της ε, Προεδρίας. Έχουμε τον κατάλογο με ό,τι ε, έχει φτάσει στα χέρια μέχρι σήμερα και σας έχουμε μοιράσει. Όποιος ενδιαφέρεται να μιλήσει με τη γραμματεία. Θέλω όμως να ξεκινήσω με κάποιες πρόσφατες ε, εξελίξεις σε θέματα εμπορικής πολιτικής. Καταρχήν, ε, για την κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΠΟΕ. 16 με 17 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα, 13 ευρωβουλευτές παραβρέθηκαν και ήταν και άλλοι 300 από τον υπόλοιπο κόσμο όπου συνεδρίασαν στη Γενέβη, στα κεντρικά του ΠΟΕ και διοργανώθηκε ε, αυτή η συνάντηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της τη Ομάδας ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων συναντήσαμε και τον κύριο Αζεβέδο που είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ και για τα θέματα των ε, εμπορικών σχέσεων της ειρήνης, της ευημερία, όπως επίσης για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον αυτές, αυτής της οργάνωσης, όπως επίσης και τους μελλοντικούς γύρους διαπραγματεύσεων. Συναντηθήκαμε με τους πρέπει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΙΠΑ και πρέπει να σας πω πως εγκρίναμε και ένα τελικό έγγραφο από το οποίο ε, το συμπεράσμα είναι πως ε, θα προσπαθήσει η κοινοβουλευτική συνέλευση να πιέσει τον, ε, τα διάφορα μέρη έτσι ώστε να καταλήξει ο γύρος της Ντόχα και να υπάρχουν όλα τα στοιχεία από το πακέτο στο Μπαλί. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία η επόμενη συνεδρίαση είναι η 34η ε, συνεδρίαση της ε, Διευθυντικής ε, Επιτροπής που θα συνεδριάσει του χρόνου του Δεκέμβριο. Εάν κάποιος που ήταν στη Γενέβη θέλει να σχολιάσει, θα χαρώ να του δώσω το λόγο. Κύριε Σούλτς, ήσασταν εκεί. Ποιος άλλος. Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι, δεν χρειάζεται να λάβετε το λόγο, συνάδελφε. Δύο σύντομα σχόλια. Καταρχήν, έχετε απόλυτο δίκαιο, ήταν πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση και θα ήθελα να τονίσω πως παρόλο που δεν συμμετείχα αυτή τη φορά στη συνεδρίαση της Steering Committee, που έγινε την προηγούμενη από την κοινοβουλευτική διάσκεψη να σας πω πως όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να επιστήσουν την προσοχή ε, μας στο γεγονός πως οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι πιο ορατοί και να παρακολουθούν πιο στενά τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΟΕ και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δίδει ιδιαίτερη σημασία πάντα στο να διατηρείται το πολυμερές αυτό σύστημα εμπορικών σχέσεων και πρέπει να στηρίξω και εγώ αυτή την προσέγγιση ε, εμείς ως ε, ίντα θα πρέπει να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωση που έχουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτό κρύβεται και πίσω από τις συζητήσεις που έγιναν και στην κοινοβουλευτική αυτή διάσκεψη και θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως ε, υπάρχει το σλόγγαν που λέει πως θα πρέπει το εμπόριο να προωθήσει την ευημερία, την ειρήνη και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε όλα τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ και αυτό εξαρτάται από την μεγαλύτερη συμμετοχή της συντεταγμένης κοινωνίας και των ε, κοινοβουλευτικών της εκπροσώπων ε, σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν κάναμε άλλο ένα βήμα έτσι ώστε να ενισχύσουμε ε, το πολυμερές αυτό σύστημα για να παραμείνει εν ζωή και για να για να προετοιμάσουμε και την Υπουργική Συνδιάσκεψη, μια και εμείς είμαστε ο σε Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα. Ε, με συγχωρείτε, θα μιλήσω για ένα άλλο θέμα, για την προτιμησιακή ε, σχέση που έχουμε με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στα πλαίσια της διάσκεψης του Μπάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 15 μέλη του ΠΟΕ είπαν πριν από δύο εβδομάδες πως θα δώσουν σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μια προτιμουσιακή ε, πρόσβαση στο χώρο των υπηρεσιών μαζί με μέτρα ε, οικοδόμησης δυναμικού και πρέπει να συγχαρώ αλλήλους για την πρόοδο Να σας πω πως ο τέταρτος ε, γύρος πραγματεύσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα τελείωσε 30 Ιανουαρίου και έχουμε τα ε, προϊόντα καθαρής ενέργειας, ΑΠΕ και ενεργειακή, ενεργειακό ανεφοδιασμό που ήταν τα θέματα. Το 2015 και το Ισραήλ και θα γίνει και μία συνάντηση ακόμα τέλη Μαρτίου. Αύριο θα ακούσουμε την παρουσίαση που θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Για τη γενική ε, συμφωνία για τις, υπηρεσίες, για τις υπηρεσίες, η ΤΙΖΑ, 9 με 13 Φεβρουαρίου συνεδριάσαμε στη Γενέβη με πολύ βαριά ημερήσια διάταξη να καλύψουμε όλα τα θέματα υπηρεσιών που καλύπτει αυτή η συμφωνία. 23 συμμετέχοντες ε, και έχουμε καινούριο κράτος στην Ουρουάη. 13 με 17 Απριλίου είναι η επόμενη συνεδρία και μία πρώτη ε, συνεδρίαση πολιτική τον Ιούλιο για να κάνουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση που γίνεται στα ε, μέσα της διαδρομής. Η ΙΝΤΑ θα οργανώσει μια μεγάλη ακρόαση για τη συμφωνία αυτή και θα συμμετέχουν και πολλοί γνωστοί εμπειρογνώμονες. Επόμενη ανακοίνωση επενδυτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μιανμά. Η συνάντηση έγινε 9 με 12 Φεβρουαρίου στη Ραγκούν της Μιανμάρ και η συνεδρία σε αυτή ήταν μια ευκαιρία για να παρουσιάσουμε στους βερμανού εταίρους μας μια πρόταση κειμένου το οποίο έχει παγιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να προστατεύονται οι επενδύσεις και μια συμφωνία που την έχει επενδυ... Ε, διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει μια διμερή συμφωνία προστασίας επενδύσεων με τη χώρα αυτή. Η Επιτροπή Ίντα θα θυμόσαστε είχε οργανώσει μια δημόσια ακρόαση ε, το Δεκέμβριο του 2014 για το θέμα αυτό αυτό είχαν έρθει οι διαπραγματευτές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας να μας μιλήσουν. Επόμενη συνάντηση το Μάιο. Τελείωσα λοιπόν με τις ανακοινώσει και έχω ένα ε, τελευταίο θέμα. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε ένα νέο υπάλληλο, τον κύριο κάβριελ Άλβαρες, που βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Ε, καλωσορίσατε στην ε, Επιτροπή μας. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Θέλετε κάτι, κυρία Πρόεδρε, μία παρατήρηση. Η τσεχική τηλεόραση βρίσκεται εκτός ηθούσης και αν το επιτρέψετε μπορεί να μπει και να γυρίσει κάποια πλάνα. Θα ήθελα λοιπόν να τους καλέσουμε, αλλά βεβαίως εξαρτάται από τη δική σας έγκριση. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από τους συναδέλφους, θα ήθελα να τους επιτρέψουμε να περάσουν. Αν οι συνάδελφοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, βεβαίως μπορούν να μπουν. Κυρία Πρόεδρε, εγώ έχω πάντα την εντύπωση πως αυτές είναι οι δημόσιες συναντήσεις, ε, οι οποίες βγαίνουν και με web stream, δεν είμαστε δηλαδή και κλεισμένων των θυρών, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ε, σαφές αυτό και το λέω για να το γνωρίζουμε και για το μέλλον. Όλες αυτές είναι δημόσιες συνεδριάσεις που κάνουμε. Ακριβώς. Παρόλα αυτά, είναι θέμα σεβασμού να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε την άδεια των συναδέλφων πριν μπει μια τηλεοπτική κάμερα. Βεβαίω, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Περνάμε στο σημείο 4 λοιπόν τη ημερήσεω διάταξη. Είναι λοιπόν για τα μεταλλεύματα που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και ψηλού κινδύνου. Το Δεκέμβριο έγινε και μια δημόσια ακρόαση. Είχαμε κάνει και μια συνάντηση πριν για να τα συζητήσουμε. Να σας πω πως η διάσκεψη των Προέδρων είπε πως είναι υπέρ του να είναι υπεύθυνη η δική μας Επιτροπή, γιατί είχαμε κάποια σύγκρουση, αν θέλετε, αρμοδιότητες με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πάντως οι εισηγητές ε, οι εισηγητέ από την Επιτροπή αυτή θα ε, είναι πάντα παρόντες και θα ενημερώνται κατά τη διάρκεια της δικής μας δράσης. Να σας πω λοιπόν πως για την έκθεση αυτή θα τη βρείτε στο φάκελό σας και έχουμε εδώ τον συνάδελφο ο οποίος θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ σωστά είπε η Αντιπρόεδρος. Έχουν ήδη γίνει δύο συναντήσεις για το θέμα αυτό για το φάκελο για, την, για το ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης ε, ε, των μεταλλευμάτων έτσι ώστε να σπάσουμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ αυτών των μεταλλευμάτων και ε, των περιοχών συγκρούσεων και ψηλού κινδύνου και εδώ είπαμε πως θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση που θα αποτελείται από τρία στοιχεία. Η νομοθεσία που συζητάμε το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτό που θα βρείτε στην κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Εξωτερικής Υπηρεσίας Δράσης και τα συνοδευτικά μέτρα για την ε, δράση αυτή και έχουμε και το τρίτο σκέλος που είναι οι διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται μέσω της εξωτερικής υπηρεσίας δράσης, μέσω του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε μέσω αναπτυξιακής ε, πολιτικής να, ε, κάνουμε, ε, να φέρουμε κάποια αποτελέσματα. Το συζητάμε στην Ίντα, ένα από τα τρία αυτά σκέλη και αυτό είναι το εμπορικό, δηλαδή η εμπορική νομοθεσία για την οποία εμείς λάβαμε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. I uh, uh, had uh, many big number of meetings with various stakeholders. Έκανα πολλές συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και εκτός Κοινοβουλίου ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ενώσεις της ε, βιομηχανίας, ενώσει πολιτών, ενώσει εκκλησιών και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητέ και όλους τους συναδέλφου στι διάφορε επιτροπέ του Κοινοβουλίου, δηλαδή ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ, για τι συναντήσει που κάναμε το τελευταίο εξάμεινο. Γιατί πρέπει να σα πω πω είναι έξι μήνε τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το φάκελο αυτό. Και μετά τις συναντήσεις αυτές καταλήξαμε σε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία σας παρουσιάζω εδώ ως σχέδιο έκθεσης. Εγώ στηρίζω σε μεγάλο βαθμό την πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σχέδιο νομοθεσίας και νομίζω πως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια εθελοντική προσέγγιση γιατί υπάρχουν τρόποι για να βελτιώσουμε την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα στοιχεία αυτά έχουν συμπεριληφθεί εδώ στην έκθεσή μου. Τρεις είναι οι στόχοι μου με τις τροπολογίες τις οποίες σας καταθέτω. Καταρχήν να εξασφαλίζουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής των εταιριών σε αυτό το σύστημα ε, θελούσιας αυτοπιστοποίησης. Δεύτερον να είναι πιο, αποδοτικός, πιο αποδοτική η νομοθεσία. Και τρίτον να υπάρχει η πραγματική συμμετοχή και έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να είμαστε παρόντες και να μας ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής προσπάθειας και κατόπιν σε όλα τα στάδια εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Το υψηλό επίπεδο συμμετοχής θα, θα επιτευχθεί με ε, βελτίωση του ορισμού του εισαγωγέα. Θα πρέπει ο ορισμός αυτός να αναφέρεται και σε πράκτορες όπως επίσης και της εταιρεία ε, ε, στο όνομα της οποίας γίνεται η τελωνιακή διασάφηση. Επίσης, ε, μεγαλύτερη συμμετοχή εισαγωγέων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τα κατάλληλα κίνητρα. Ο κανονισμός θα πρέπει να παρέχει περισσότερη ορατότητα στις προσπάθειες των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κατάλογο υπεύθυνων εισαγωγέων που θα τον προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση μια έκθεση για την εφαρμογή ε, του κανονισμού από τα κράτη-μέλη και ο κατάλογο αυτό θα πρέπει σε τακτικά διαστήματα να ενημερώνεται. Είναι πολύ σημαντικό οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να προστατευθούν, θα ήθελα να συμπεριληφθούν και θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα, τα κατάλληλα κίνητρα, έτσι ώστε να συμμετέχουν και αυτέ στο σύστημα τούτο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να τους προσφέρουμε την κατάλληλη βοήθεια έτσι ώστε να βρεθούν και αυτές σε θέση να συμμετέχουν στο σύστημα ε, με τη δική τους επιχειρηματική λογική. Θα πρέπει δηλαδή να αποδείξουν και οι ίδιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πως είναι υπεύθυνε ε, ενώπιον των πελατών τους. Για να είναι πιο αποδοτικός δεν πρέπει να έχουμε επικάλυψη ελέγχων αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα συστήματα του κλάδου που βασίζονται όλα ε, στην οδηγία του ΟΣΑ για την δέουσα επιμέλεια και αυτή τη στιγμή αποδίδουν καρπό. Άρα λοιπόν τα σύστημα, σύστηματα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ισοδύναμα μετά από το σύστημα αυτοπιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια μέσα σε ένα πολύ στενό και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, τη στιγμή δηλαδή εισαγωγής της νομοθεσίας. Έχουμε επίσης και κάποια μέσα τα οποία έχουν στηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα την οδηγία για την υποβολή αναφορών για μη χρηματοπιστωτικά θέματα και αυτό το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις να αναφέρουν ε, τι έχουν κάνει στο θέμα αυτό της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού μιλήσαμε με τον ΣΑΟ, όπως επίσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι θα πρέπει να εισάγουμε και μια μεταβατική περίοδο έτσι ώστε το σύστημα να ε, λειτουργήσει σωστά από την αρχή. Η μεταβατική αυτή περίοδος είναι απαραίτητη για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τοποθετήσουν και αυτά, να στήσουν μάλλον ένα σύστημα πιστοποίησης και για να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως και τα 28 συστήματα ε, πιστοποίησης, τα κράτη-μέλη ε, λειτουργούν έτσι ώστε να μην ε, μπορεί κάποια εταιρεία να γυρίζει από κράτος σε κράτος και να επιλέγει το σύστημα αυτοπιστοποίησης που τη βολεύει καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε και αυτή η δική μου πρόταση μια μεταβατική περίοδο δύο ετών και μετά τα πρώτα δύο χρόνια πλήρους εφαρμογής να γίνει μια αναθεώρηση και μετά κάθε τρίτη χρονιά όχι κάθε έκτη, όπως προτείνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κάθε τρίτη χρονιά να γίνεται κάτι αντίστοιχο. Για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει έλεγχος και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό που προτείνω είναι να υπάρχουν κάποιες πρακτικές ε, ε, ε λύσεις, για παράδειγμα ομάδες επιρρογνωμόνων που θα ε, συνεδριάζουν για συγκεκριμένα θέματα με την παρουσία των δικών μας εκπροσώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, θα παρουσιάσει μια καθηγητήρια γραμμή για την ενιαία ε, εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές και τις εθνικές αρχές. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα το αφήσω εδώ. Μια τελευταία μόνο παρατήρηση. Κάναμε διάλογο και με τις πολιτικές ομάδες και με τους σκιώδες ηγητές στην Ίντα και το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου και του γεγονότος πως ακόμα και στην Επιτροπή Ντέβε αλλά και στην Επιτροπή Άφετ έχουν ήδη ετοιμάσει πολλές τροπολογίες για τις γνωμοδοτήσεις που θα ψηφιστούν και θα παρουσιαστούν ε, σε εμάς. Προτείνουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο διαφέρει κάπως από το αρχικό. Προτείνουμε λοιπόν στην Ίντα να δούμε τις τροπολογίες στις 18 Μαρτίου και να ψηφιστούν στην Ίντα ε, κατά την συνάντησή μας του Απριλίου, δηλαδή στις 13 Απριλίου τρέχοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητάς ή εισηγητρίας. Η κυρία Αρένα, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε εισηγητά για την ανάπτυξη του θέματος και την έκθεση. Να επανέλθουμε στον πρωταρχικό στόχο της πρωτοβουλίας, της νομοθεσίας δηλαδή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχει θετικό αποτέλεσμα για επίλυση του αρχικού προβλήματος, δηλαδή τη διακοπή δηλαδή της συνδέσεως μεταξύ του εφοδιασμού ε, πρώτων υλών και της περιοχής συγκρούσεων. Αυτό ήταν και το πρώτο κίνητο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη βάση μελετών των ΗΕ άλλωστε αποκαταστάθηκε ένα σύνδεσμος μεταξύ του εφοδιασμού της χρηματο... δηλαδή πρώτων υλών, της χρηματοδότησης ένοπλων ομάδων σε συγκεκριμένες περιοχές κύβου στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό αλλά βεβαίως όχι μόνο αυτή και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει ωστόσο ως υπόδειγμα για το εγχείρημα που κάνουμε. Εδώ δεν χρειαζόμαστε νομοθετήματα για να ε, εξασφαλίσουμε την καλή συνείδηση της Ευρώπης. Αντίθετα, χρειαζόμαστε μια νομοθεσία που να είναι αποτελεσματική όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή εφοδιασμό σε πρώτε και συγκρούσεις, αλλά και να μπορεί και να εφαρμοστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τελικό ωφελούμενο, που δεν είναι η ευρωπαϊκή βιομηχανία για μένα, αλλά ο πελάτη. Δηλαδή αυτό ο οποίο τελικά θα αγοράσει το προϊόν και αυτός θα, θα θέλει να είναι βέβαιος ότι το προϊόν, το τελικό προϊόν που αγοράζει είναι φτιαγμένο με τρόπο υπεύθυνο. Έχει έρθει, έχουν έρθει πρώτες ύλε από χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά, αλλά θέλει να ξέρει τι ακριβώς αγοράζει εδώ στην Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι διασκέδασα, βέβαια δεν είναι διασκεδαστικό, με την ανάλυση τριών υποθέσεων εργασίας. Η πρώτη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να δούμε δηλαδή τι γίνεται μέσα στις ροές μιας ε, προσέγγισης μόνο για τα ανάντι και τι συμβαίνει στις αγορές. Δηλαδή βλέπετε από τη μια μεριά τι συμβαίνει στη διαφάνεια δηλαδή στις χώρες προέλευσης, ορυχεία, ε, τοπικοί διαπραγματευτές, διεθνείς διαπραγματευτές. Εκεί δεν μπορεί κανείς βέβαια να κάνει τίποτε. Εκεί έχουν, ε, έχουν κάνει τις ρυθμίσεις τους. Βλέπετε στο upstream έχουμε τις, ε, τα μεταλλουργία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού εκείνους αφενός οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν υπεύθυνα και όλους τους υπολείπους οι οποίοι δεν ε, προσεγγίζουν το θέμα υπεύθυνα. Έχουμε τα μεταλλουργία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού εκτός ευρωπαϊκού συστήματος, τα τελευταία δηλαδή, κάτω δεξιά στην ε, διαφάνεια που είναι 95% σήμερα και σύμφωνα με την υπόθεση της Κομισιόν θα βρείτε ένα, μια αγορά του υπολείπου όπου η Κομισιόν δεν θα οθήσει αυτούς που είναι από κάτω από τη γραμμή να πάνε από πάνω. Βλέπετε από την άλλη μεριά όλα αυτά τα βέλη εφοδιασμού των διαφόρων συνιστοσών και των τελικών προϊόντων στα κατάντη που επιτρέπονται από τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει απολύτως καμία διαδικασία στα κατάντη, στο downstream δηλαδή. Αυτός που παράγει ένα αριθμό ε, προϊόντων που συναποτελούν τελικό προϊόν δεν έχει κανένα κίνητρο για να ε, επιλέξει μια υπεύθυνη προσέγγιση. Δηλαδή που αγοράσει οτιδήποτε από οπουδήποτε. Αυτό δεν προτείνει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Δεν πρόκειται να τροποποιήσει τις συμπεριφορές αυτές. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αγορά Μεταλλουργίων και Εξευγενιστών θα παραμείνει εξαιρετικά περιορισμένη, μάλιστα και θα εξαφανιστεί στο βαθμό όπου κοστίζει λιγότερο να πάνε να εφοδιαστούν από αλλού, να τροφοδοτηθούν από αλλού, όπου οι τιμές δεν καθορίζονται από το τι κάνει κανείς καλά ή όχι, αλλά από τη θέση έχει στην διεθνή αγορά. Είτε ακολουθεί υπεύθυνη πολιτική είτε όχι, η τιμή είναι ίδια. Και αν περάσουμε τώρα από την πλευρά των βιομηχανιών, τότε εφόσον οι τιμές δεν ποικίλουν σύμφωνα με την προσέγγιση που έχετε, τότε πάτε να προμηθευτείτε εκεί που οι τιμές είναι φτηνότερες. Και εφόσον ο λιανέμπορος που είναι ο πελάτης σας δεν έχει καμία ε, διαφάνεια μπροστά του, επομένως δεν ξέρει πού μπορεί, πού αγοράζει. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση που μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι τέτοια που να μπορέσει να αλλάξει τα όσα βρίσκονται από την άλλη μεριά, στα νάντι δηλαδή στις χώρες προέλευσης δεν θα προστατεύσει ούτε και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, αντίθετα, θα υποκατασταθούν σε αυτές αλλοδαπές επιχειρήσεις και τελικά ο Ευρωπαίος πελάτης δεν θα γνωρίζει τι, ποιο είναι το τελικό προϊόν που αγοράζει. Και επομένως θα ωφεληθεί τελικά η μη υπεύθυνη προσέγγιση στα προϊόντα που δεν είναι ευρωπαϊκά. Αυτή λοιπόν η υπόθεση εργασία δεν εκπληρώνει κανένα στόχο. Ούτε στην πρώτη φάση, α πούμε, ούτε στο κέντρο, ούτε στη δεύτερη φάση. Έρχομαι σε μια δεύτερη υπόθεση και όπως ο κύριος Βίνκλερ είπε, συναντηθήκαμε με πολλού ενδιαφερομένους. Εκεί λοιπόν εξέτασα μια μεικτή υπόθεση. Ε, μια ρύθμιση υποχρεωτική στα νάντι και μια ε, εθελοντική στα κατάντι. Τι θα οδηγήσει, τι θα οδηγήσει αυτό, είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η διαφάνεια αυτή που θα δείτε τώρα από την προηγούμενη, αλλά πάλι δεν ευνοεί την υπεύθυνη στάση με την έννοια ότι όπως έλεγα πριν τα μη ευρωπαϊκά μεταλλουργία ανέρχονται στο 95% της αγοράς και δεν θα έχουν κανένα ιδιαίτερο συμφέρον ε, να λάβουν τα μέτρα αυτά της δέουσας επιμέλειας γιατί ο τελικός καταναλωτής θα έχει την επιλογή ανάμεσα σε δύο προϊόντα είτε το υπεύθυνο προϊόν είτε το μη υπεύθυνο προϊόν. Στην περίπτωση πάλι αυτή η αγορά δεν λειτουργεί για να επιβάλλει τις ρυθμίσεις αυτές. Δεν οδηγούμεθα λοιπόν προς μια υπεύθυνη προσέγγιση και θα έχουμε πάντοτε μια συμβίωση του ανεύθυνου και του υπεύθυνου με κυρίαρχη θέση του ανεύθυνου. Πάλι το αποτέλεσμα εκεί είναι μικρότερο σε ό,τι αφού δηλαδή του αρχικού στόχου. Και έχουμε και την τρίτη υπόθεση εργασίας που αυτή βασίζεται στον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων σε όλη την αλυσίδα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Από κάτω μέχρι πίσω, δηλαδή προς τα πάνω. Εκεί βλέπετε και μια διευκρίνηση του ποιος είναι, διευκρίνηση υπέρ μάλλον του τελικού ε, πελάτη, του τελικού αγοραστή, αλλά ξεκαθαρίζουμε και την ευρωπαϊκή αγορά και για, τα μεταλλουργία και για τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού και για τη βιομηχανία και αυτό μας ενδιαφέρει όλες και όλους να έχουμε αποτελεσματικές και υπεύθυνε επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα όχι μια προσέγγιση που θα είναι υποχρεωτική σε όλη την αλυσίδα και επιτυγχάνει τον πρώτο στόχο που είναι μια υπεύθυνη προσέγγιση μέχρι τη χώρα προέλευσης, αλλά και μια εγγύηση για το ότι τελικά η βιομηχανία μας θα κερδίσετε από αυτό. Εξηγώ λοιπόν έτσι σύντομα για ποιο λόγο η υποχρεωτική προσέγγιση σε όλη την αλυσίδα δεν θα ενοχλήσει το βιομηχανικό σύστημα, αλλά αντίθετα θα εξασφαλίσει ώστε η Ευρώπη να διαθέτει μια βιομηχανία που να είναι δυνατόν να τροφοδοτεί και τους πελάτες της με υπεύθυνα προϊόντα, και ταυτόχρονα να μπορέσει να επηρεάσει και στις ε, περιοχές συγκρούσεων μέσω μιας διαδικασίας υπεύθυνου εμπορίου. Στο όνομα λοιπόν της ομάδας μου θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια αλλά λαμβάνουν υπόψη και την ανάγκη συνοδείας των επιχειρήσεων αυτών. Όπως είπε ο κ. Βίνκλερ πριν είναι σημαντικό να υπάρξει και μια περίοδος προσαρμογής για την εφαρμογή του συστήματος και θα είναι ενδιαφέρον λοιπόν να υπάρχουν και κάποιες μεταβατικές περίοδοι για την εφαρμογή του συστήματος και βέβαια να ληφθεί υπόψη και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και θα δείτε ότι όσο πηγαίνετε προς το downstream, δηλαδή προς το τελικό προϊόν, τόσο πιο πολύ τίθεται, πιο έντονα δηλαδή, τίθεται το θέμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που χρειάζονται λοιπόν καθαρά συνοδευτικά μέτρα για ε, την υποχρέωση αυτή, που είναι και υποχρέωση που απορρέει από το κώδικα του ΩΣΑ. Θα καταθέσουμε λοιπόν αυτές τις ε, τροπολογίες που δεν επιτρέπουν συμβίωση των συστημάτων όπως αυτή προβλέπει ο κ. στην έκθεση του ΔΕΗ και το σύστημα του ΩΣΑ και το σύστημα των ε, επιχειρήσεων. Είναι ένα σύστημα στο οποίο συμμετέχουν 151 χώρες του ΩΣΑ, 151 χώρες και θέλουμε αυτή η μοναδική παραπομπή που κάνουμε να είναι στον ΩΣΑ και όχι στις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει ορισμένες, ορισμένοι βιομηχανικοί όμιλοι. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα διατυπώσουμε τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε και ελπίζουμε έτσι να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία που να είναι θετική και για τις χώρες προέλευσης και βεβαίως να λαμβάνει υπόψη και την ευρωπαϊκή κατάσταση, την οικονομική ευρωπαϊκή κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Αρενά. για τους ECR, Σαντέρο Λόμες. Ευχαριστώ να μου επιτρέψετε να μιλήσω Ολλανδικά κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Κλάρκ κολλείεται δυστυχώς διότι υποχρεώται να παρίσταται σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Ευχαρίστω όμως να λάβω εγώ το λόγο εκ μέρου τη, Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολλή δουλειά που έχει ήδη κάνει για το σημαντικό αυτό θέμα το οποίο αγγίζει πολλούς ανθρώπους. Έχουμε ακούσει ήδη πολλές απόψεις. Όλοι ωστόσο, λίγο πολύ, επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Θέλουμε δηλαδή να διακοπεί η χρηματοδότηση ενόπλων συγκρούσεων μέσω της εμπορίας αυτών των προϊόντων που συχνά εξορίσονται με παράνομο τρόπο ή ε, γίνονται αντικείμενο παράνομη εμπορίας κλπ. Η έκθεση πετυχαίνει να διατηρήσει μια ισορροπία. Η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, αντίθετα με τα όσα ακούσαμε μόλις πριν από την κυρία συνάδελφο, προτιμά να διατηρηθεί η προσέγγιση του εισηγητού και να δοθεί περισσότερη προσοχή στην παροχή κινήτρων προς την κατεύθυνση αυτών δεν κινηθούν οι διάφοροι οργανισμοί για τη θέσπιση ενός συστήματος ευθύνης, για παράδειγμα με την ε, κατάσταση ενός καταλόγου υπεύθυνων παραγωγών. Και έχω τώρα και ορισμένα επιμέρους σχόλια. Όπως είπε και ο κ. Βίνκλερ, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπτύξουμε νέα συστήματα. Έχουμε κανόνες για την δέουσα επιμέλεια και για την καθαρή αλυσίδα προμηθειών που έχει θεσπίσει ο ίδιος ο κλάδος, ο οποίος έχει λάβει μέτρα, για παράδειγμα στην ε, αγορά χρυσού του Λονδίνου. Να μην υπάρξει όμως επικάλυψη των προδιαγραφών, των στάνταρτ, να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι κανόνες, να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές προσαρμογές έτσι ώστε να αποφύγουμε και την υπερβολική γραφειοκρατία. Σημαντικό κυρίως είναι, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθούν κίνητρα και κυρίως να καταστρωθεί ένας κατάλογος ηλεγμένων, υπεύθυνων προμηθευτών και εισαγωγέων. Εξάλλου η πίεση των ομοτήμων, αυτό το peer pressure, είναι πολύ σημαντικό και πολύ ισχυρή η πίεση αυτή η οποία επιτυγχάνει να αποδώσει αποτελέσματα. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να φτιάξουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, για την παράγραφο 7β που γίνεται παραπομπή σε συστήματα δέουσας προσοχής του κλάδου. Υπάρχουν τέτοια συστήματα, υπάρχουν τέτοια, τέτοιες ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη. Γι' αυτό εδώ εκφράζουμε μια επιφύλαξη. Δεν θα πρέπει να είμαστε και ανοιχτοί απέναντι σε ενδεχόμενες καινοτόμες προτάσεις που μπορούμε να συμπεριλάβουμε και να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Να ασκήσουμε δηλαδή κάποια πίεση και μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ίσως να μπορέσει να επιτευχθεί καλύτερα αυτό με ε, καινοτόμους κανόνες στο μέλλον. Τώρα, ε, τρίτο, ανακυκλωμένα υλικά. Εκεί η ομάδα μου, η πολιτική μου ομάδα, δηλώνει ικανοποιημένη που προτείνεται ένα φιλόδοξο αλλά λογικό σύστημα. Εμείς διαθέτουμε επαφές με τον κλάδο και έχουμε κατανοήσει ότι απαιτείται μια ρεαλιστική προσέγγιση. Γιατί αλλιώς καθίσταται σχεδόν αδύνατο να διαπιστωθεί η προέλευση των ορυκτών. Εκεί το καλύτερο είναι να τηρηθούν οι κανόνες του ΟΟΣΑ. Αυτό επιθυμούμε να περιληφθεί ρητά μάλιστα στην ε, πρόταση κανονισμού. Ε, μας ικανοποιεί επίσης η διετής μεταβατική περίοδος που προτείνει ο εισηγητής. Το μόνο ερώτημα που τίθεται εδώ είναι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε τακτικότερη ενημέρωση, τακτικότερες αναφορές, γιατί αυτό ταιριάζει καλύτερα με τις απαιτήσει μας. Να έχουμε τακτικότερες αναφορές εκθέσεις και τακτικότερους ελέγχους για την επίτευξη των ε, επιθυμητών αποτελεσμάτων. Και το τελευταίο σχόλιο μου κάτι το οποίο είχε θέσει η συναδελφός μου, την οποία εκπροσωπώ σήμερα. Το σχέδιο εκθέσεως βασίζεται σε ένα σύστημα όπου η εποπτική αρχή συνυποστηρίζεται από τις 28 χώρες μέλη. Εμείς, ωστόσο, σκεπτόμαστε ότι ίσως είναι καλύτερο να υπάρχει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος να ασκεί την εποπτεία με τρόπον ώστε να εγγυάται μια ενιαία εποπτεία και να αποφεύγονται και οι επικαλυπτόμενες γραφειοκρατικές και βέβαια και οικονομικές επιβαρύνσεις. Ευχαριστώ πάντως και πάλι τον εισηγητή και αναμένω την παραπέρα καρποφόρο συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Φιλελεύθερη, κυρία Δεσσαρδέζ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια βεβαίω κύριε Σιγητά, πολύ καλή δουλειά. Το κείμενό σας ενισχύει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί καλή βάση για την παραπέρα εργασία μας. Βέβαια, να μην χάσουμε από τα μάτια μας όλες και όλοι εδώ ότι στόχος του κανονισμού θα πρέπει να είναι να σπάσει αυτή η διασύνδεση μεταξύ των ορυκτών, της εξόριξη δηλαδή των πρώτων υλών και της χρηματοδότησης ε, ενόπλων σειράξεων. Βεβαίω και χρειάζεται μια ρεαλιστική προσέγγιση, χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο είναι αποτελεσματικό, να μην μειώνει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μα και ταυτόχρονα να επιτρέπει να διεξάγεται ο αγώνα κατά αυτή τη διασύνθεση θα εξετάσουμε τον μηχανισμό που την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ίσω να ισχύσει και ω μοντέλο και για τον υπόλοιπο κόσμο και να επιτρέψει την ανάπτυξη μια θετική δυναμική, έτσι ώστε και άλλε χώρε να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Οι χώρε ε, τη περιοχή των ε, μεγάλων λιμνών στην Αφρική, αλλά και η Κίνα έχουν αρχίσει να κάνουν βήματα προ την κατεύθυνση αυτή. Τάση η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί. Το βλέπουμε ήδη από την αρχή της συζητήσεώς μας ότι τίθεται ένα μέγα ερώτημα για τον χαρακτήρα εθελοντικό ή δεσμευτικό του συστήματος. Εθελοντικό ή υποχρεωτικό. Διάβασα, συζήτησα, προβληματίστηκα πολύ. Δεν έχω καμιά προκαθορισμένη ιδεολογική τοποθέτηση για το θέμα αυτό. Νομίζω εν τέλει όμως ότι θα πρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία να λάβει χαρακτήρα δεσμευτικό. Όχι σε όλο το οικονομικό πεδίο, θα πρέπει ωστόσο να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αναγκαστικό χαρακτήρα τουλάχιστον για τα μεταλλουργία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού τα ευρωπαϊκά υπενθυμίζω άλλωστε απηχώ εδώ βέβαια και τον δόκτωρα Ντενί Μουκεμπέ ο οποίος ε, έχει τιμηθεί με το βραβείο Ζαχάρο φέτος για τον αγώνα κατά των ενόπλων Σημαντικό μήνυμα λοιπόν ο δεσμευτικός χαρακτήρας τουλάχιστον για τους βασικότερους ε, παίκτες εντός εισαγωγικών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε παραπέρα. Δεν θέλουμε να μειωθεί και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας που ούτως ή άλλως έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα ε, τελευταία. Βεβαίως και πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα κινούνται προ την κατεύθυνση αυτή, προς την άσκηση της δέουσας επιμέλεια, δηλαδή. Χρειάζεται άρα μια κατάλληλα επιλεγμένη προσέγγιση και οι επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να συμμορφωθούν με τα συστήματα δέουσας επιμέλεια, να επωφεληθούν γιατί όχι από μια σήμανση που θα χορηγεί η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και να πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εξασφαλίζει την ποιότητα της αλυσίδας προμηθειάς της. Έτσι ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να εμπιστευτεί την σήμανση αυτή. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι άλλοι μικρότεροι επιχειρηματίες γενικά να μπορέσουν να αναλάβουν τις πρωτοβουλίε και όσοι αναλάβουν τις πρωτοβουλίε, να έχουν την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. για να λειτουργήσει το σύστημα. Άρα ένα ξεκάθαρο υποχρεωτικό μήνυμα προς τους μεγάλους βασικούς φορείς της αλυσίδας αυτής, αλλά και ένα ξεκάθαρο κίνητρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι νομίζω ότι είναι το καλύτερο να προχωρήσουμε. Ακούγοντάς σας όλες και όλους βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί κάποιος λογικός συμβασμός. Και ο δρόμος προτείνω νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Για να ολοκληρώσω, να μην λησμονούμε ότι ό,τι και αν θεσπίσουμε από μόνο του δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των ορυκτών που προέρχονται από χώρες όπου σημειώνονται σειράξει. Αλλά χρειάζεται και μια πολιτική, μια εξωτερική πολιτική και μια διπλωματική πολιτική λογική η οποία να μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ όλους και όλους. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πάντα θετική του προσέγγιση. Ο κ. Σόλτς. Ενωτική Αριστερά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την σκληρή του δουλειά. Όπως ήδη είπε, είχαμε διάφορες συνεδριάσεις και συζητήσεις για αυτό το σημαντικό θέμα. Διοργάνωσε λοιπόν αυτές τις ανταλλαγές απόψεων και συναντήσεις και το εκτιμώ. Να είμαι ειλικρινής. Ο φάκελος αυτός που αφορά τα μεταλλεύματα είναι από τους πιο σημαντικούς που πρέπει να εξετάσουμε κατά τη διάρκεια τη θητείας μας. Αφορά όλη την πενταετία και είναι ένα οριζόντιο θέμα. Αφορά συγκρούσει, σειράξει, διαπραγματεύσει που δεν έχουμε ολοκληρώσει. Είναι μια πρόκληση λοιπόν. Υπάρχουν και υπήρξαν πάρα πολλοί πόλεμοι για φυσικού πόρου. Πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι και παιδιά επίσης υποφέρουν από τη σκλαβιά και πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε την ειρήνη είχαμε και πρόσφατα την κοινοβουλευτική συνέλευση που το υπογράμμισε αυτό και υπάρχουν προσδοκίες για την Ένωση ως εταίρο για το σύστημα αυτό να συμβάλλει συμβαστικά και καθοριστικά σε αυτή την πρόκληση. Και όπως είπαμε προηγουμένως απονείμουν το γραφείο Σαχάροφ σε έναν μαχητή για αυτά τα θέματα. Και συμφώνησαν οι Υπουργοί από 43 ε, χώρες για την ύπαρξη μιας διαδικασίας ΕΛΕΚ όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού και τη διαδικασία της. Και αυτό βεβαίω περιγράφεται στον οδηγό τη δεύτερη επιμέλεια. Και θα έλεγα ότι όλε οι κυβερνήσει με διάφορα κόμματα που τι αποτελούν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν για μια νέα διαδικασία και δεν βλέπω γιατί να μην μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για μια νομοθεσία ώστε να θεσπιστούν τελικά προδιαγραφές όσα. Εγώ βέβαια θα το υποστηρίξω αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και τι απαραίτητε τροπολογίε. Νομίζω ότι οι ιδέε είναι καλέ του εισηγητή, θα ήθελα όμω να προσθεθούν και κάποια άλλα ζητήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά ώστε να ακολουθήσουμε τι επιθυμίε των πολιτών μα στην Ένωση, που θέλουν να βεβαιωθούν ότι δεν χρηματοδοτούμε σε πράξει και πολέμους έστω και αν συγκεντρώμαστε σε κάποια επιμέρους αιτήματα και έχουμε εμπειρία τέλο πάντων για κάποιες διεθνείς πτυχές ε, αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις μας να ανταποκριθούν σε αυτά τα αιτήματα και θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισοδυναμία για όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό το θέμα οριζόντια σε όλη τη διάρκεια της αλυσίδας. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ρυθμιστικό υποχρεωτικό. Θα πρέπει να επεκτείνουμε και την ομάδα των επιχειρήσεων, να τη διευρύνουμε. Θα πρέπει να δίνουμε βεβαίως και τη δυνατότητα να υπάρχει παρέκκληση όπου είναι απαραίτητο και θα πρέπει ε, τα συνοδευτικά μέτρα να υποστηρίξουν αυτή την νομοθεσία ώστε να υπάρχει ανάπτυξη Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι προς τους αυτούς μας, προς τα κοινοβουλία και προς τους πολίτες. Και νομίζω περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται απλά και μόνο γενικά και αόριστα για το τι θέλουμε, αλλά έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία οφείλονται σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Η ομάδα μου λοιπόν υποστηρίζει όλες τις τροπολογίες οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη αυτού του στόχου και θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μου για άλλη μια φορά να υπάρχει λογική από όλε τι ομάδε στην Επιτροπή μα και ελπίζω στην ολομέλειά μα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και Σουρτ. Η κυρία Μοργαντίνη. Σαρχεντίνη, όχι Μοργαντίνη. Η κυρία Μοργαντίνη έχει έτσι μια θέση που την καλοβλέπω, αλλά ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί. Με συγχωρείτε λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σκακελέο δεν είναι εδώ στις Βρυξέλλες σήμερα. Μου ζήτησε να την αντικαταστήσω, κάτι το οποίο θα πράξω. Και το εκτιμώ. Στη συζήτηση που κάναμε για πάνω από έξι μήνες, από το καλοκαίρι, μάλλον πάνω από 4,5 χρόνια, από το 10, το καλοκαίρι του 10, όπου είχε εξεγγίσει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία και υπήρχε παρανόηση για το τι ακριβώς σημαίνει δέωσα επιμέλεια και το τι ακριβώς σημαίνει κατευθυντές γραμμές για, για τα μεταλλεύματα από τον ΩΣΑ. Δέωσα επιμέλεια αποτελεί νομίζω ακριβώς την ε, διαδικασία η οποία αφορά την ακρίβεια των δηλώσεων. Το γεγονός ότι εμείς συζητάμε το κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή θελούσε αυτό. Νομίζω ότι ακριβώς ενισχύει τους φόβους που υπάρχουν γιατί οι προτάσεις από τον ΩΣΑ αφορούν ακριβώς αυτή τη δέουσα επιμέλεια και τις κατευθυντήριες γραμμές για το εμπόριο. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις καθ' όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τους πιο μικρούς στους πιο μεγάλους και τους βοηθάμε να εφαρμόσουν την νομοθεσία και να βελτιωθούν. Γι' αυτό ακριβώ η πρόταση του εισηγητή για καθυστέρηση και να ε, υπάρχει διετία μεταβατική τι να σα πω, όλο το εγχείρημα αυτό είναι μεταβατικό γιατί στην ουσία δεν σταματά την εισαγωγή μεταλλευμάτων όταν είναι μεταλλεύματα που έρχονται από περιοχή σειράξεων λέμε ότι εντάξει τα δεχόμαστε και σιγά σιγά θα βελτιώσουμε την διαφάνεια στην ε, λυσίδα φοδιασμού. Γι' αυτό ακριβώ και η Κομισιόν στις προτάσεις της που βασίστηκαν έτσι πολύ ελαφρά, πάρα πολύ ελαφρά όμως στις καθε, καθε, γραμμές του ΩΣΑ θα έκανα ακόμα πιο αόριστα όλα αυτά. Υπάρχουν όμως αυτές οι κατευθύνσεις γραμμές της δεύτερης επιμέλειας από το ΩΣΑ που υπογράφηκαν από όλα τα μέλη του και από ό,τι ξέρω και από, όλες τις, από όλα τα μέλη όλες τις χώρες της Ένωσης και τις χώρες της περιοχής των μεγάλων λιμνών με μια διαδικασία όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι, μικροί, μεγάλοι, η επιχειρηματική κοινότητα κτλ. όλοι συμμετείχαν. Έχουμε επίση μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του τι συμμόρφωση κάνουμε όταν είμαστε ένας μεγάλος όμιλος πολυεθνικός και, μια, και άλλο το τι κάνουμε όταν είμαστε μια μικρομεσαία το γεγονό ότι οι μικρομεσαίε δεν μπορούν να συμμορφωθούν, αυτό αντιμετωπίζεται από τι κατευθύνσει γραμμέ του ΩΣΑ. Αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι που δεν το, ότι δεν διευκολύνουμε του εαυτού μα να πάμε πίσω δηλαδή στι αρχικέ κατευθύνσει γραμμέ του ΩΣΑ, να το κοιτάξουμε και να το κάνουμε νομοθεσία. Το είπε και ο Χέλμου προηγουμένω. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσαμε αυτό που είπε και η κυρία Μαρία Ρένα προηγουμένω, δηλαδή το πώ να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ μα επιχειρήσει δεν θα επιδιδών, δεν θα χειροτερεύουν επειδή θα πρέπει να εφαρμόζουν νομοθεσία που άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν. Οπότε αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα ήταν επιδερμικό, δηλαδή επιλεκτικά διαλέγουμε κατευθυντήριες γραμμές και περιζόμαστε στην διαφάνεια, στα χιτήρια, αλλά δεν δίνουμε στα χιτήρια κίνητρα ώστε να κάνουν το σωστό, ώστε να μην ε, φτάσουμε τελικά στο αρχείο. Εμείς οι πράσινοι προτείνουμε τροπολογίες όσον αφορά την κατεύθυνση του υποχρεωτικού. Δηλαδή να πούμε ότι αυτή η δοσοπημελία είναι ήδη υποχρεωτική. Ένα είδος ήπιας νομοθεσίας, ήπιου δικαίου. Όσον αφορά δηλαδή την παραγωγή αγαθών και οτιδήποτε προέρχεται από χιτήρια ή οτιδήποτε ας πούμε προέρχεται από την νοτιοανατολική Κίνα δεν θα ελέγχεται και η Ευρωπαίοι από από πού ε, έρχονται αυτά τα προϊόντα. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα εμπορεύματα άνθρακα στην Κολομβία, συγκεκριμένα μεταλλμάτα από την Μιανμάρ και το γεγονό ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν περιορίζεται στην περιοχή των μεγάλων λιμνών είναι θετικό. Όμως, όμως, θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλα εμπορεύματα τα οποία οδηγούν σε βία και σειράξεις. Είμαι πεπισμένη ο, ότι ο πρώην Επίτροπος για το Εθνές Εμπόριο Ντεχούχτ ήθελα να αντιμετωπίσω το θέμα της σειράξης στο Κονγκό μέσω πρότασης που θα αντιμετώπιζε το θέμα του εμπορίου των μεταλλευμάτων, αλλά δεν πήγε αρκετά μακριά. Δεν κατέστησε μια πρόταση που να κάνει τη διαφορά. Οπότε ή θα το κάνουμε σωστά τώρα ή δεν θα το κάνουμε καθόλου. Αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα δεν θα έχει αντίκτυπο στο Κονγκό και αλλού. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει εμείς να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Πεκίνο από το Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή, τον συνάδελφο, για αυτή τη δύσκολη δουλειά που έκανε. Και τον ευχαριστώ επειδή συνέταξε μια βασική πρόταση που μπορούμε να συμμεριστούμε. Να υπενθυμίσω πάντως ότι το εμπόριο φυσικών πόρων βρίσκεται πίσω από τις, κάποιες από τις πιο βίαιες σειράξεις στον κόσμο και στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είμαστε υπεύθυνοι κι εμείς γι' αυτό είμαι στη υπεύθυνη για την βοήθεια σε ενόπλες ομάδες, την επιμήκυση των πολέμων, υπεύθυνη επειδή είμαστε διάφοροι για την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ευρώπη είναι μια από τις κυριότερες αγορές εξαγωγών πολλών φυσικών πόρων και πάρα πολλούς από αυτούς τους πόρους που δέρχονται από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ελερωμένες με αίμα. Γι' αυτό ακριβώς αυτό που κάνουμε εδώ θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μαζί με άλλους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένω και εγώ είμαι υπέρ ενό υποχρεωτικού συστήματο που θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλου τους φυσικούς πόρους αντικείμενο εμπορίου, εμπορίου που οδηγεί σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται χρονικά και να εφαρμόζει διάφορου πόρου μέσω και ευέλικτων νομοθετικών εργαλείων όπω τις κατεξουσιοδοτήσει πράξη. Και με του αδέλφου μου θα ήθελα να υιοθετήσουμε μια δέσμη κανόνων βασισμένους στους κανόνες του ΩΣΑ που θα ε, ε, επιβάλλουν αντίστοιχους κανόνες και σωστούς κανόνες στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, κυρίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι όλο και περισσότερο διότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί απαιτούν την απόδειξη οι φυσικοί πόροι να προέρχονται από εμπόριο που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε εξαιρούν, εξαιρούν τις μικρομεσαίες, τις εξαιρούν όμως και από τους μεγάλους δημοσίου διαγωνισμού. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα να υπάρχει ισορροπία. Η αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ στην κοινωνία των πολιτών αυτών των χωρών που μα ζήτησαν να θεσπίσουμε δίκαιου κανόνε που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να ρυθμίζουμε μια και καλή το εμπόριο αυτών των μεταλλευμάτων και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο το Κοινοβούλιο πρόθεσε αυτέ τι αρχέ με ένα ψήφισμα για τι εμπορικέ Πρακτικέ που είναι υπεύθυνε και που υιοθετήθηκε πριν από ένα έτο. Νομίζω λοιπόν έφτασε η ώρα να τηρήσουμε τι υποσχέσει μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιγκίν. Τελειώσαμε με τους Κιώδης. Μπουτιχόφερ και Μεταμέ λείπουν. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους Μορέλ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι για τους στόχους, ότι πρώτον, καταρχάς δεν μπορούμε να θαρρύνουμε το εμπόριο εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, συμφωνούμε όλοι για το γεγονό ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε το ότι εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μεταφράζεται σε σειράξεις που καταστρέφουν χώρες ολόκληρες. Τρίτο, συμφωνούμε όλοι νομίζω για το ότι θα πρέπει να προωθήσουμε στο και δεν εύκολο το ηθικό εμπόριο και τέταρτον στην πεποίθησή μας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επιθυμούν και θέλουν να γνωρίζουν από πού έρχονται αυτά τα προϊόντα, την αυσιμότητα Μετά λοιπόν την σημερινή συζήτηση και όπως η κυρία Ρένα θεωρώ και εγώ ότι καλώς υπάρχει ο τωρινός κανονισμός αλλά του λείπει φιλοδοξία και δυστυχώ, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι αποτελεσματικό. Επειδή το κυριότερο πρόβλημα είναι κατά πόσο εμεί ε, θέλουμε ή μπορεί κανεί να προσχωρήσει σε αυτόν τον εθελούσιο χαρακτήρα ή όχι. Το, το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό ακριβώ και οδηγεί σε στρεβλώσει μεταξύ αυτών λοιπόν που θέλουν να είναι υπεύθυνοι και αυτών που δεν το επιθυμούν. Και τελικά αντιμετωπίζετε το ίδιο και οι δύο. Και αυτό που κάνουμε λοιπόν, να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο δεν είναι αποτελεσματικό. Οπότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτή την έννοια τη αυτοπιστοποίηση τη εθελοντική με την υποχρεωτική πιστοποίηση. Οι υποχρεώσει ε, να αφορούν όλη την αλυσίδα παραγωγή. Και μετά το ρεαλιστικό ζήτημα που τίθεται είναι το πώ θα συνοδεύσουμε, πώ θα βοηθήσουμε τι επιχειρήσει, ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες. Αυτό πρέπει να μα απασχολήσει σήμερα και νομίζω ότι είναι πιθανό να θέσουμε ένα χρονοδιάγραμμα και το εφαρμόσουμε. Αν όμως εγκαταλείψουμε την έννοια ή το νόημα του υποχρεωτικού χαρακτήρα, αυτά που θα κάνουμε θα είναι αποτελεσματικά και θα μου το αντίθετο αποτέλεσμα. Και μάλιστα δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση, αλλά αναφέρεται νομίζω στι τροπολογίε. Εγώ αναρωτιέμαι κατά πόσο το πεδίο που καλύπτει ο κανονισμό για του φυσικοπόρου, πόρου αν αρκεί. Γιατί συνέχεια υπάρχουν και άλλα μεταλλεύματα και άλλα ορυκτά και άλλοι πόροι που είναι αντικείμενο σειράξεων σε διάφορε χώρε. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά στη συζήτηση για τι τροπολογίε. Πάντω, καλώ όλου του συναδέλφου να εξετάσουν το κατά πόσο δεν παρακάμπτουμε ακριβώ το στόχο μα, αν δεν κάνουμε το σύστημα αυτό υποχρεωτικό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Σφαϊνά. Είναι πάντα ωραίο να έχει κανείς τέτοιου είδους νομοθετικές προσπάθειες που όλοι συμφωνούν στο ποιος είναι ο στόχος και όλοι θέλουν να κάνουν το σωστό. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το σωστό και πώς θα το πετύχουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την εξής σκέψη πως το εμπόριο με τα, για τα αγαθά αυτά είναι πολύ σημαντικό για τις πιο φτωχές χώρες και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι φτωχές αυτές χώρες θα μπορούν να συνεχίσουν να εμπορεύονται τα αγαθά αυτά ε, προς όφελος της ευημερία τους και της μάχης που δίνουν για να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Δεν θα πρέπει δηλαδή να καταφέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή το εμπόριο να στηρίξει τον λαθασμένο στόχο και να ωφεληθούν οι λάθος άνθρωποι και όχι οι σωστοί. Εδώ λοιπόν είναι το βασικό ερώτημα και νομίζω ότι ο τρόπος που θα μας επιτρέψει να το πετύχουμε είναι να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι απλό. Εγώ στο ΕΛΚ ήμουν υπεύθυνο ε, στην γνωμοδότηση για την ξυλία όπου προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της λαθροϊλοτομίας και ξέρετε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόβλημα με την περίπλοκη νομοθεσία. Μπορεί και να την προτιμούν, γιατί βέβαια αυτό δυσκολεύει πιο πολύ τις μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό αποτελεί και ένα φραγμό για την είσοδο των νέους στον κλάδο. Οπότε κάποιες εταιρείε που φέρνουν ανάπτυξη στις φτωχές χώρες μπορεί να είναι μικρές, μπορεί να είναι εγχώρια, συμβέλεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει το σύστημα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό γίνεται. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κοίταξαμε πολύ ενδιαφέρον ε, τα διάφορα σχεδιαγράμματα που παρουσίασε η κυρία Ρένα. Δεν μπορώ να πω πως τα κατάλαβα όλα. Όμως δεν είμαι σίγουρος γιατί η τελευταία εικόνα που μας δείξατε μοιάζει να είναι πιο απλή. Ως διαφάνεια τουλάχιστον. Αλλά δεν είμαι σίγουρος πως την πραγματικότητα για τους ε, εμπορευόμενους θα είναι και τους φορείς θα είναι ε, η πιο απλή λύση. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κρίνουμε και επανέρχομαι στην ε, νομοθεσία για την ξυλία. Εκεί καταφέρουμε πολλά, πολλά σωστά, κάποια λάθη. Η μεγάλη πρόκληση είναι η εξής. Όσο πιο περίπλοκο είναι το σύστημα που στείλουμε, το, τόσο, πιο δυσκολεύουμε, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουμε την εφαρμογή και τον έλεγχο. Ξέρουμε λοιπόν πως αυτοί οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τους κανόνες και να κάνουν το σωστό είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν τους κανόνες είτε είναι υποχρεωτικό είτε όχι. Οπότε, αν το σύστημα είναι τόσο περίπλοκο που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε παρκώς, τότε θα κυνηγάμε τελικά αυτούς οι οποίοι δεν νοιάζονται να εφαρμόσουν. Αυτή είναι η βασική αλήθεια και θεωρώ πως η πρόταση και του κυρίου Βίγκλερ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ισορροπημένες. Και κάθε νέα τροπολογία που έχουμε από τους σύγητες θα πρέπει να εξεταστεί αλλά υπό αυτό το πρίσμα θα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα ή πιο απλά γιατί αν όντως απλουστεύει το σύστημα τότε θα το βελτιώσει κιόλα. Και τέλος, υλικά ανακυκλώσιμα. Κανείς δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα, αλλά πολλοί συνάδελφοι σε άλλες εκθέσεις έχουν ζητήσει να ενταχθεί αυτό το σκέλος. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω να μην το κάνετε, γιατί καταρχήν αυτό είναι ο χώρος στον οποίο συνήθως δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και δεύτερον, νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στο μέλλον έτσι κι αλλιώς πρέπει να το προωθήσουμε και θα πρέπει να κάνουμε τον κλάδο αυτό πιο ανταγωνιστικό, πώς βοηθώντας τον να απαλλαγεί από οποιαδήποτε δύσκολη και περίπλοκη νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλος που θέλει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτό το σχέδιο έκθεσης, όπως επίσης και την ευκαιρία να συνεισφέρει στις σημερινές σας συζητήσεις για τα διάφορα στοιχεία τα οποία θίξατε ως Επιτροπή. Ποια είναι η θέση μας. Νομίζω ξεκαθαρίσαμε στο σχέδιο κανονισμού το ότι η πρότασή μας βασίζεται στα εξής στοιχεία και θα τα επαναλάβω. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να προωθήσουμε μία υπεύθυνη ε, μια υπεύθυνη πορεία ε, στην ε, εξοχή μετάλλων από περιοχές υψηλού κινδύνου και να ακολουθήσουμε μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και γι' αυτό επιλέξαμε και την επωνομαζόμενη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό να επιτευχθεί μέσω όλων των κοινοτικών πολιτικών και μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας που προσφέρουν, αλλά και μέσω της διπλωματικής οδού. Τα βασικά αυτά στοιχεία αναφέρονται και στην ανακοίνωση της ΥΠΑ της της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και όταν μιλάμε για μέταλλα από περιοχές σύγκρουσης θα πρέπει αυτό που θα προκρίνουμε είναι μια ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υπεύθυνα μέταλλα, που θα βελτιώσει και την κατάσταση επιτόπου. Η προσέγγιση μας αυτή και για να προωθήσουμε την εισαγωγή ε, βολφραμίου, τανταλίου, χρυσού και κασίτερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την εισαγωγή των μετάλλων που εξορίχθηκαν και τυχαν επεξεργασίας με υπεύθυνο τρόπο προτείναμε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Η λογική που κρύβεται πίσω από αυτή την προσέγγιση ακολουθεί τις βασικές αρχές. Δηλαδή, στοχευμένη και γι' αυτό αναφερόμαστε στα βασικά σημεία της αλυσίδας ανεφοδιασμού, τα χιτήρια καταρχήν, γιατί μετά το χιτήριο είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς ποια είναι η πηγή ενός μεταλλεύματος ή ενός ορυκτού και είναι αναλογική η προσέγγιση μας γιατί υπάρχει αυτή η εθελούσια ε, πλευρά η οποία βασίζεται στα κίνητρα που θα δώσουμε έτσι ώστε να μην φέρουμε και κάποιο αρνητικό αντίκτυπο για τις περιοχές σύγκρουσης και είναι και ε, η οποία στοχεύει ανάντι και όχι κατάντι ε, αντίθετα με το όσο κάνει σχετική νομοθεσία των ΙΠΑ που μέχρι στιγμής ήταν μάλλον ανεπιτυχής και θα έλεγα και επιζήμια για τις χώρες παραγωγούς. Μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από την εμπειρία μας, γιατί έχουμε και τον κανονισμό για την ξυλία που ήδη αναφέρθηκε στην αίθουσα και δεν νομίζω πως χρειάζεται να επαναλάβω ποια είναι τα λάθη τα οποία εντοπίσαμε να κάνουν οι άλλοι. Η προτινόμενη αυτή νομοθεσία αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο, αλλά δεν θα δώσει την τελική λύση, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα, όλες τις επιπλοκές και το περίπλοκο του ζητήματος. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω τη σημασία που έχουν τα μέτρα που θα λάβουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις Ξέρω πως αρκετά, αρκετοί ευρωβουλευτές ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί και θα παρακολουθεί τα προτινόμενα μέτρα και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά. Δηλαδή, εντοπίσαμε ποια είναι τα εργαλεία που χρειάζονται έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια επιτόπου για να φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα ξεκινήσαμε και κάποιες εξουστρεφείς δράσεις με χώρες επεξεργασίας όπως η Κίνα και η Ινδία και θα εντατικοποιήσουμε και τις σχέσεις αυτές με άλλους εταίρους, οι οποίοι είναι σημαντικοί σε επίπεδο παραγωγής, κατανάλωσης ή επεξεργασίας. Θέλουμε να δούμε τέλος ποιος μπορεί να δράσει καλύτερα αυτόνομα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έτσι ώστε να κινήσουμε μια πρωτοβουλία υπόλοιπη υπεύθυνης εξόριξης και να γνωρίζουμε ακριβώς πώς προχωράει το θέμα και να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι για οποιασδήποτε αλλαγές. Τέλος, αλλά εξίσου σοβαρό είναι τα κίνητρα, το είπατε κι εσείς. Δηλαδή να δούμε και το θέμα κατάντι, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές προμήθειες. Αποτελούν και τα θέματα και, αυτά τα θέματα τμήμα της δικής μας ανακοίνωσης όπως επίσης και το πώς θα επηρεαστούν από τα προγράμματα αυτά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταγράφω τις προτάσεις που παρουσιάσετε και βεβαίως θα εξετάσω τα θέματα αυτά ε, με πολλές λεπτομέρειες και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ τώρα Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπατε κι εσείς, είναι όντως ένας κανονισμός και ένα θέμα το οποίο είναι πολύ τεχνικά, αλλά και παράλληλα βαθιά πολιτικά. Άρα λοιπόν χρειάζομαι πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι έχω στη διάθεσή μου για να δώσω μια απάντηση στις προτάσεις που μου υποβάλλατε. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να δώσω ε, κάποιες απαντήσεις. Ελπίζω η Μαρία Ρένα, η εξωτερική συνάδελφος, να μην το πάρει προσωπικά, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα του ανταγωνισμού και της τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Γιατί ε, και γελάστε μαζί μου. Λοιπόν, μόνο τις δικές σας διαφάνειες είδαμε συνάδελφε. Σβήστε τα σας παρακαλώ και με συγχωρείτε αν το αστείο μου δεν ήταν και τόσο αστείο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Για τα τεχνικά ζητήματα. Είπατε πως πρότεινα να καθυστερήσει δύο χρόνια να τεθεί σε εφαρμογή. Όχι. Οι συζητήσεις που έγιναν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο με οδήγησαν στο να προτείνω μία εισαγωγική περίοδο ε, διετή γιατί χρειάζεται να οικοδομήσουμε το σύστημα με τον τρόπο που επιλέγουμε. Δεν είναι καθυστέρηση λοιπόν, είναι περίοδος προετοιμασίας εισαγωγής του συστήματος. Τώρα για μια ενιαία ευρωπαϊκή αρχή να περάσουμε στο πολιτικά ευαίσθητο αυτό θέμα. Γιατί μια αρχή θα ήταν μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά βιώσιμο. Όταν όλοι μιλάνε για λιγότερη γραφειοκρατία, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιπροεδρία για την απλούστευση της νομοθεσίας, να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πούμε εμείς ότι χρειάζεται να στήσετε μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία, ακόμα και αν είναι εξαιρετικός ο στόχος που επιδιώκεται, νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα απορριφθεί και δεν κρίνω πως είναι βιώσιμη. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς μια νέα ευρωπαϊκή αρχή να την προτείνουμε πολλές προτάσεις έγιναν για την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα αυτού του κανονισμού. Και εγώ έχω δεσμευθεί ε, στο να συνεισφέρω σε έναν τέτοιο αποτελεσματικό κανονισμό. Όμως, αποτελεσματικός κανονισμός αυτός είναι αυτός που είναι εφαρμόσιμος. Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο κανονισμός δεν θα λειτουργήσει στην πράξη. Όπως είπε και ο Κρίστοφερ, μας έδωσε το παράδειγμα της λαθροϊλοτομίας. Μπορούμε εμείς με κανονισμό να απαγορεύσουμε την λαθρό Αλλά τι αποτέλεσμα θα φέρει, θα σταματήσει την λαθροϊλοτομία Όχι, άρα λοιπόν εφαρμόσιμους κανονισμούς, εφαρμόσιμη νομοθεσία. Αρκετοί συνάδελφοι είπαν πως θα πρέπει να διδαχθούμε από τη δική μας εμπορία αλλά και την εμπειρία άλλων. Διαπιστώνω και το βλέπετε κι εσείς πως η σχετική νομοθεσία τον είπα είναι πραγματικά αμφιλεγόμενη και τα αποτελέσματά της είναι αμφιλεγόμενα και δεν έχουμε κάποια συνενετική άποψη για το πώς λειτουργήσε στην πράξη αυτή η νομοθεσία. Άρα λοιπόν αυτό το δίδαγμα θα, το πρέπει, θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Το τι θα, πώς θα λειτουργήσει η πίεση του Ευρωπαίου καταναλωτή και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, το peer pressure. Εδώ νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι η εκπαίδευση. Ξέρω πως δεν ικανοποιούν τους συναδέλφους τα ισοδύναμα συστήματα. Δηλαδή έχουμε τα διάφορα προγράμματα για την υπεύθυνη εμπορία μετάλλων, για τα υπεύθυνα χιτήρια κτλ. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Αν πούμε σε κάποιους από τους εμπλεκόμενους, από τους φορείς οι οποίοι ήδη έχουν στήσει και συμμετέχουν σε ε, κάποιες ε, προσπάθειες υπεύθυνης ε, αν τους πούμε πολύ ωραία όλα αυτά που κάνατε αλλά ξέρετε εμείς δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και θα πρέπει να ξεκινήσετε πάλι εκ του μηδενός. Δεν νομίζω ότι αυτό ε, θα έχει θετικό αντίκτυπο και τέλος επειδή δεν έχω πια άλλο χρόνο στη διάθεσή μου πρέπει να σας πω και δεχτείτε το αυτό, είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου. Και όταν υπάρχει μεγάλη συνένεση στην πολιτική, πολλοί λένε πως δεν θα συμβεί τίποτα. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας, φαντάζομαι πως ισχύει το αντίθετο και θα είναι πολύ καλή νομοθεσία που θα προκύψει από αυτές μας τις συζητήσεις. Κάνατε πολύ καλή δουλειά συνάδελφοι, είναι δύσκολο το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι. Επόμενη συζήτηση τροπολογιών 18 και 19 Μαρτίου στην Ίντα. 13-14 Απριλίου στη συνάντησή μας θα ψηφίσουμε και μετά θα περάσει από την Ολομέλεια στις 18 με 21 Μαΐου. Άρα λοιπόν θα γίνουν κάποιες συναντήσεις με ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα είχαμε το χρόνο να ανταλλάξουμε απόψεις και θεωρώ πως είναι σημαντικό. Ίσως δεν ήταν η στιγμή της συνένεσης, αλλά νομίζω ότι και ο συμβιβασμός θα βρεθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Είναι το σχέδιο έκθεσης για την μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία. Ο κύριος Λαντσμπέργκης είναι ο εισηγητής. Βρίσκεται στο φάκελό σας και αυτή η έκθεση και μια και είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Δύο εκπροσώπους της Κομισιόν έχουμε σήμερα εδώ, ο κύριος Γκρίσο και ο κύριος Λιβεντάλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. αξιότιμα μέλη της ΙΝΤΑ, θα ήθελα καταρχήν να σας ενημερώσω για το πώς έχει οικονομική κατάσταση στην Ουκρανία. Ξέρετε κι εσείς πως η κατάσταση έχει χειροτερεύσει πολύ σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη επιχείρηση μακροοικονομικής στήριξης που εγκρίθηκε. Έχει, έχουμε τις συνεχιζόμενες σειράξεις στα ανατολικά της χώρας με αποτέλεσμα μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι οικονομικές μεταβλητές χειροτερεύουν συνέχεια ε, και από την εποχή που υπεγράφει το πρώτο πρόγραμμα με το Δουνουτού τον Απρίλιο. Η ύφεση είναι πολύ πιο βαθιά και συνεχιζόμενη από ό,τι είχε ε, από είχαμε προβλέψει, 7,5% έπεσε το ΑΕΠ, ενώ το πρόγραμμα του Δουνουτού είχε προβλέψει 5% πτώση και συνεχίζεται ε, η πτώση του ΑΕΠ ε, με γοργούς ρυθμούς γύρω στο 15% ανατρίμηνο και ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2015 όπου ξέρουμε πως 21% ήταν η αιτήσια μείωση στη βιομηχανική παραγωγή. Άρα λοιπόν το ΔΝΤ και ε, ε, οι εθνικές αρχές πιστεύουν πως και φέτος θα παίξει τουλάχιστον 5% το ΑΕΠ φέτος. Το νόμισμα ε, υποτιμήθηκε πολύ σημαντικά τα αποθέματα συναλλάγματος έχουν συρρυκνωθεί. 50% έχασε πέρσι το νόμισμα και άλλα 25% φέτος μέχρι τώρα το Φεβρουάριο. Τα αποθέματα έχουν χάσει το 60% πέρσι των αποθεμάτων των συλλαγματικών πέρυσι και τον περασμένο μήνα επίσης πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν έχουν μόνο 6,4 δις ε, στη διάθεσή τους, το οποίο καλύπτει ένα μήνα εισαγωγών οι ενεργειακές ταρίφες ε, που μεταβλήθηκαν έφεραν τον πληθωρισμό πολύ πιο ψηλά από ό,τι είχε προβλέψει το πρόγραμμα του Δουνουτού με αιτήσιο προϋπολογισμό το 28, κάτι της εκατό ε, ήταν η αύξηση μέχρι φέτος. Το έλλειμμα είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, όχι γιατί η κεντρική κυβέρνηση ε, κάνει δαπάνες, γιατί είναι πολύ σφιχτή η πολιτική της, αλλά η μεγάλη εταιρεία τους αερίου ε, και πετρελαίου ε, έχει μειώσει ε, τον όγκο εργασίας κατά τουλάχιστον 10% πέρσι με αντίστοιχη μείωση της συνεισφοράς της εταιρείας αυτής στο ΑΕΠ της χώρας. Ξέρετε πως πάρα πολλές τράπεζες επίσης χρειάστηκαν να κλείσουν ή έχουν μπει σε διαδικασία πτώχευσης. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σκοτεινή η εικόνα η οποία επηρεάζεται και από τις πολιτικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει και μεγάλη αβεβαιότητα γιατί θα γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Το, οι διεθνείς δωρητές λοιπόν ε, υπό την ε, σκέπη του Δουνουτού ξαναυπολόγησαν τις ανάγκες χρηματοδότησης για τα επόμενα δύο χρόνια, αυξήθηκαν αυτές και έχουν ένα νέο πακέτο στήριξης το οποίο αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται, επαναλαμβάνω με βασική ε, πρωταγωνιστικό ρόλο του δονουτού, έτσι ώστε να υπάρχει ένας πιο ε, μακρύς χρηματοδοτικός μηχανισμός στήριξης μέχρι το 2017 τουλάχιστον ε, και έχουμε και άλλους δωρητές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα με στόχο μία αναδιάρθρωση ε, του δανείου που βρίσκεται στα χέρια του ιδιωτικού κλάδου. Ε, άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο στις 8 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτό το νέο σύστημα ε, μακροπιστωτικής στήριξης για ένα ποσό 1,8 δις μετά από δύο πολύ ευαίσθητε επιχειρήσει που κάναμε, που ήταν συνολικό προπολογισμό στο 1,6 δι, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ήδη αποδεσμευθεί, μένει απλώ μια τελευταία δόση 250 εκατομμυρίων. Και εδώ πρέπει να δούμε αν σέβονται την αιρεσιμότητα για να μπορέσουμε να το εκταμιεύσουμε και αυτό. Ξέρετε πω αυτή είναι η μεγαλύτερη τέτοιου είδου στήριξη που έχουμε προσφέρει και πρέπει να σα πω ότι αν συγκριθεί με προηγούμενε, θα φτάσουμε σε ποσά τα οποία δεν έχουμε γνωρίσει ε, το ποσοστό. Επίσης έχουμε ε, και ένα δάνειο γύρω στα 300 ε, εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουμε. Άρα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης από, χώρα Ευρωπαϊκής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρα που δεν είναι μέλος της. Και η συνδρομή αυτή θα είναι με τη μορφή δανείων όπως είχαμε και στο παρελθόν, με μία σειρά προϋποθέσεων έγκρισης, όπως όλα τα ε, προγράμματα θα πρέπει να δέχεται τα πολιτικά προαπαιτούμενα, δηλαδή δημοκρατικοί θεσμοί, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και δεύτερον, σε στενό συντονισμό με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που έχει υποβάλει εκθέσεις και θα τις βρείτε στην εκ των προτέρων αξιολόγηση των προτάσεων θα πρέπει να εξετάσουμε και το ρεκόρ ε, και τα επίπεδα εφαρμογής και την υπόδοση σε ε, εφαρμογή του προγράμματος του προηγούμενου με το Δούνου του με την ε, παράλληλη με τον παράλληλο σεβασμό τη ερεσιμότητας που υπάρχει στο μνημόνιο που έχει υπογράψει η χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε να οικοδομήσουμε στη βάση των προηγούμενων χώρων στους και κλάδων στου οποίου έχουν γίνει μεταρρυθμιστικέ προσπάθειε, σύμφωνα με τι 75 προτεραιότητε που έχουν ε, τοποθετήσει οι διεθνεί θεσμοί, μάχη κατά τη διαφορά, φορολογική διοίκηση, ενδυνάμωση του περιβάλλοντος επενδύσεων, ε, κλαδικέ και ε, μεταρρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλει να υπογραμμίσει πόσο σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα. Τρέχει ο χρόνος και πιέζει αφόρητα. Ξέρετε κι εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να ακολουθήσει την ε, νομοθετική διαδικασία. Ακούμε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Ξέρετε για την προηγούμενη ε, προσπάθεια που έγινε, που ενέκριναν ε, οι συνομοθέτες, το ένα δις πήγε υπό την ε, έκτακτη διαδικασία άρθρο 213, δηλαδή μία απόφαση του Συμβουλίου χωρίς επίσημη έγκριση από πλευράς Κοινοβουλίου, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και επίγουσα, εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως έχουμε την δειγμένη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυρίζουμε, επιστρέφουμε στην τακτική μας νομοθετική διαδικασία. Όμως, στείλαμε επιστολές στην Προεδρία του Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Ίντα πως θα πρέπει να επιταχύνουμε πιέζει ο χρόνος γιατί οι μεγάλες ε, ε, ανάγκες, ε, τις, οι χρηματικές ανάγκες της Ουκρανίας συγκεντρώνονται στο 2015. Άρα λοιπόν στο σχέδιο που έχουμε, αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και έχουμε έγκριση από τους συνομοθέτες, θα πρέπει η πρώτη δόση να πληρωθεί πριν το καλοκαίρι, μια δεύτερη δόση πριν τα τέλη του χρόνου και μια τρίτη δόση το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Οποιαδήποτε επιπλοκή στη διαδικασία έγκρισης μπορεί να μας καθυστερήσει με την πρώτη δόση και να ξεπεράσουμε το χρόνο, ορίζοντα το χρονικό του ε, καλοκαιριού. Εμείς δεν μπορούμε ε, να χρηματοδοτήσουμε στη μέση του καλοκαιριού και καταλαβαίνετε πως λόγω των μηνυμάτων που μας έχει στείλει το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε όλα αυτά να γίνουν μέχρι το καλοκαίρι. 3 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο ε, ε, είπε πως θα στείλει μια πρόταση χωρίς τροπολογία στην Κορεπέρ έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα ε, δράσουμε ταχύτητα και ελπίζουμε πως το ίδιο θα κάνει και το Κοινοβούλιο. Η Κορεπέρ συμφώνησε σε αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να παροτρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης έτσι ώστε οι προτάσεις αυτές να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν. Ε, χωρίς τροπολογίες, για παράδειγμα, όπως πρότεινε ο εισηγητής. Και ιδανικά αυτό να γίνει στην Ολομέλεια με πρώτη ανάγνωση στις 25 Μαρτίου. Η πρόταση αυτή σέβεται απόλυτα τις ε, αρχές που έχουμε για τις μακροοικονομικές δράσεις που στις 12 Αυγούστου συμφωνήσαμε. Άρα λοιπόν το κείμενο είναι πραγματικά πανομοιότυπο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τις προηγούμενες αποφάσεις. Ελπίζω πως αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διαδικασία λήψη απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να σας δώσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται και να σας συνδράμει όσο μπορείτε για να επιταχύνουμε με τη διαδικασία αυτή. Merci. Euh, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή, κύριο Λαντσμπέργκης. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η μακροοικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι πολύ σημαντική. Ιδίως σε περίοδο συστημικών οικονομικών προβλημάτων και βαθιάς ύφεσης που έχει κληρονομήσει η νυν Ουκρανική κυβέρνηση. Θα ήθελα πρώτα να τονίσω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει μόνη της. Η διεθνής κοινότητα συμμετέχει στην ε, υποστήριξη προς την Ουκρανία. Όταν μιλούμε για Ουκρανία βλέπουμε εικόνες καταστροφής. Βαριά ρωσικά μηχανήματα ή βαριά με ρωσικά ε, άρματα περνούν από ουκρανικές πόλεις και το καθεξής περνάει δύσκολου καιρού η Ουκρανία. Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα για να εκπληρώσει τι υποχρεώσει που έχει αναλάβει με τη Συμφωνία Συνδέσεω είναι και οι ίδιε μια σημαντική πρόκληση. Αλλά πρέπει να τα κάνουν αυτά. Λίγοι πιστεύουν ότι η εκεχηρία θα κρατήσει με το ρόλο που παίζει η Ρωσία βέβαια. Μετά από συναντήσεις με άλλους συναδέλφους άλλων πολιτικών ομάδων φαίνεται καταρχήν να υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Βεβαίω είναι και στρατηγική σημασία του θέματος αλλά και επίγονο χαρακτήρας του. Σήμερα βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τη μεγαλύτερη στην ιστορία της α, οικονομική υποστήριξη προς μια χώρα που δεν αποτελεί μέλος της και βέβαια και δεν αρκεί. Χρειάζονται όμως οι διαδικασίες διότι προβλέπονται τρεις δόσεις 600 εκατομμυρίων ήδη φέτο δύο από αυτέ. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει η πρόταση αυτή χωρί τροπολογίε και όσο γίνεται γρηγορότερα για να διασφαλίσουμε ώστε η πρώτη δόση να φτάσει στην Ουκρανία ήδη στι αρχέ του καλοκαιριού. Ήδη το Συμβούλιο Υπουργών έχει δώσει την καταρχή συμφωνία του για να προχωρήσει χωρί τροπολογίε. Αυτό λοιπόν μπορεί να το πετύχει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Εξωτερικών ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. πιο σχεδιασμένη ωστόσο προσέγγιση και λιγότερο ad hoc. Ελπίζω λοιπόν ότι και το Συμβούλιο θα εγκρίνει το σχετικό ψήφισμα για περαιτέρω υποστήριξη προς την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ αγαπητέ κύριε. Οι πολιτικές ομάδες και οι οδησηγητές για τους Σοσιαλιστέ και δημοκράτες, ο κύριος Βοστινάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι μόνο μου άρεσαν οι δύο τοποθετήσει που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τον εισηγητή κ. Μπέργκη. αλλά εγώ θα προσθέσω και λίγε παρατηρήσει για να βοηθήσω να κατανοήσετε όλοι και όλε την έκτακτη, τον έκτακτο χαρακτήρα της κατάστασης στην Ουκρανία αλλά και των στρατηγικών μας σχέσεων με την Ουκρανία. Ουκρανία δεν είναι υπόθεση business as usual. Χρειάζεται να μην λησμονούμε ότι γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Και κάθε μέρα ο πόλεμος αυτός κοστίζει από 5 έως 7 εκατομμύρια την ημέρα. Αυτό είναι το κόστος του πολέμου αυτού που επιβλήθηκε στην Ουκρανία. Όχι επειδή το ήθελε. Δεύτερο, μεταξύ των απολειών, μην λησμονείτε ότι πέρσι η Ουκρανία όχι μόνο έχασε την εδαφική της ακερότητα αλλά έχασε και σημαντικούς οικονομικούς πόρους από την ανατολική πλευρά της χώρας που είναι τώρα εκτός κυριαρχίας της ε, ε, κεντρικής κυβέρνησης αλλά φαίνεται να είναι και εκτός πάσης εθνικής κυριαρχίας. Επιπροσθέτως δε του κόστους της μετάβασης και ούτω καθεξής. Για το λόγο αυτό ή για τους λόγους αυτούς πρέπει να χειριστούμε την συμφωνία αυτή ως κατεπίγουσα με την ελπίδα ότι ο κατεπήγον χαρακτήρας δεν θα γίνει βέβαια και ο βασικός κανόνας για όλα όσα έχουμε να κάνουμε για την Ουκρανία. Όμως στο συγκεκριμένο πλαίσιο για το οποίο μιλούμε είναι σημαντικό να γίνει τώρα να προχωρήσει η πρόταση χωρίς τροπολογίες έτσι ώστε να εγκριθεί το δυνατόν συντομότερο και γι' αυτό η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υποστηρίζει την έγκριση της προτάσεως της Κομισιόν άνευ τροπολογιών και άνευ ιεσδήποτε καθυστερήσεως έτσι ώστε να μπορέσει η πρόταση αυτή να εγκριθεί μέχρι τον Απρίλιο και να προσφερθεί στο στρατηγικό εταίρο στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα αυτό καλύπτει μόναχα ένα μέρο των στατικών σχέσεών μα με την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει και άλλα βαριά προβλήματα. Και όπω είπαν οι άλλοι συναδελφοί μου πριν, πρέπει βεβαίω να εξετάσουμε την εφαρμογή τη συμφωνία, να εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανική κυβέρνηση δαπανά ορθά τα χρήματα που τη δίνονται μέσω τη συμφωνία συνδέσεω και βεβαίω και τη μακροοικονομική υποστήριξη, Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν μέσα στα πλαίσια της διμερούς μας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας. Αυτό βεβαίως δεν αποτελεί μόνο χειρονομία αλληλεγγύη θα πούν ορισμένοι, ούτε μόνο στρατηγική ή διάσταση των σχέσεών μας με τη χώρα αυτή, μπορεί να πούν άλλοι. Αλλά είναι σημαντικό η Ευρώπη σε αυτή τη δραματική περίοδο που περνάει η χώρα να δείξει αλληλεγγύη και να της προσφέρει υποστήριξη για να την βοηθήσει να περάσει τις δραματικότερες αυτές στιγμές που έχει περάσει η περιοχή αυτού του κόσμου μετά από την πτώση των τυχών που υποτίθεται ότι άνοιξαν νέους ορίζοντες για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Κάποια μαθήματα δεν ξεχάστηκαν, αλλά κάποια άλλα ίσως, άλλα ίσως ξεχάστηκαν. Και εμείς πρέπει να διδαχτούμε βεβαίω και νέα πράγματα από την κρίση για να βελτιώσουμε στη δική μας προσέγγιση και τις σχέσεις μας με τις γειτονικές μας χώρες. Η δέσμη αυτή μέτρων αποτελεί μέρος του εργαλείου πολιτικής γειτονίας. Το κρίνουμε λοιπόν ως πολύ σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσουμε την χώρα να ξεπεράσει τις δυσκολίες της και να αποκαταστήσει τη λειτουργία μιας οικονομίας που χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη μπορεί να καταρρεύσει ή να αναγκαστεί να καταρρεύσει με ενέργειες εκείνων των αρπακτικών που επιβουλεύονται την Ουκρανία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακλάρκιν. Όχι. Δύο βουλευτές δείχνουν ένα στον άλλο. Α, όχι, δεν λοιπόν η κυρία Μακλάρκιν, ο κύριος Ζαχραντήλ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. αντικαθιστώ τον κύριο Πιέρχα που δυστυχώς κολλείεται σήμερα. Σύντομα λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο συνάδελφός μου εξ ονόματος της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών τίθεται υπέρ της προτάσεως επιθυμώ να επαναλάβω, όπως θα έλεγε και ο ίδιος, ότι η σχεδιαζόμενη στήριξη θα πρέπει να δοθεί υπομορφήν δανείου και να χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού που θα διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της Ουκρανίας, και κατά κάποιο τρόπο είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι και άρα είμαστε σχεδόν θα έλεγα υποχρεωμένοι να προσφέρουμε την στήριξη αυτή στην Ουκρανία. Και γι' αυτό συμφωνούμε με την μορφή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα με μια κίνηση των δυνατών τάχιστη. Ευχαριστώ. Εκ των φιλελευθέρων, ο κύριο Βαν Μπάλεν. Όντως είναι κατεπίγουσα κατάσταση όπως είπαν και άλλοι προηγουμένως και για τον λόγο αυτό πράγματι θέλουμε και εμείς να επιληθεί το θέμα το συντομότερο δυνατό χωρίς τροπολογίες υποστηρίζουμε στην περίπτωση αυτή λοιπόν τα όσα προτείνει ο συγητής. Το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι εξής. Βεβαίως η Ουκρανία έχει κατακομματιστεί από τη Ρωσία και από τα πρωτοπαλικαρά της και βλέπουμε ότι το Μίνσκ 2 πάει να γίνει όπως και το Μίνσκ 1. Ωστόσο η Ουκρανία πρέπει και να μεταρρυθμιστεί. Υπό τι παρούσε περιστάσει, βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει να μεταρρυθμίσει την οικονομία τη, πρέπει να θεσπίσει κράτο δικαίου και εμεί πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία όχι μόνο με παροχή χρημάτων, αλλά και στην προσπάθεια αυτή μεταρρυθμίσεων. Βεβαίω, η ομάδα μου Αλντε ευχαρίστω ε, θα ε, υποστηρίξει, αλλά έχω και τη συνάδελφό μου δίπλα μου που θα ήθελα να προσθέσει κάτι, άλλο στον επόμενο γύρο. Εσείς κύριε Σόλτς τώρα της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κατανοήσει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση της Ουκρανίας και οικονομικά και αλλιώς και ότι είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στήριξη. Όμως είναι τρίτη φορά που ασχολούμαστε με την συζήτηση της μορφής που πρέπει να λάβει η αδίποτε μακροοικονομική στήριξη προς την Ουκρανία. Ως πολιτική ομάδα την τελευταία φορά είπαμε ήδη ότι αυτή η μακροοικονομική στήριξη θα πρέπει να δοθεί υπό συγκεκριμένους όρους μεταρρυθμίσεων. Στην παράγραφο 2.2.2 του παραρτήματος της πρότασης της Κομισιόν λέει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και μέθοδοι πρέπει να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένοι. Ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί σήμερα να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα όσα έως τώρα έχει και μπορεί να επαληθεύσει ότι ανταποκρίνονται στο master plan της Γενικότερης Συμφωνίας με την Ουκρανία. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι χρειαζόμαστε την μακροοικονομική στήριξη. Όμως αυτή πρέπει να είναι αμέση απευθείας στήριξη για την ανοικοδόμηση της οικονομίας στη χώρα. Και εκεί να συζητηθούν και να θεσπιστούν μαζί με τις πολιτικές αρχές της Ουκρανίας συγκεκριμένα προγράμματα αυτά τα accompanying policy programs to be agreed with the Ukrainian authorities, ποια θα είναι. Και μιλούμε για 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται. Και έρχομαι στο κύριο ερώτημα. Από την τελευταία δόση που προβλεπόταν για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης του στρατού στην Ουκρανία, ένα τρίτο του ποσού αυτού κατέληξε σε τσέπε ιδιωτών. Δεν έφτασε ποτέ στις δομέ της χώρας. Πώ εξασφαλίζουμε σήμερα λοιπόν ότι οι επόμενες δόσεις θα καταλήξουν να δεσμευτούν υπέρ των συγκεκριμένων στοχευμένων μέτρων. Ποιο μας το εγγυάται αυτό. Και μιλούμε για χρήματα φορολογουμένων των πολιτών της Ένωσης που βεβαίως τα προσφέρουμε για αλληλεγγύη, υποστήριξη, ξεπέρασμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μια γειτονική χώρα, αλλά η προϋπόθεση πρέπει να είναι ότι αυτά θα χορηγηθούν για την κοινωνική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Αν δεν καταφέρει η Ουκρανία να σταθεροποιήσει τις εσωτερικές εξελίξεις της χώρας αυτής, να σταθεροποιήσει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να δώσουμε και άλλες δόσεις, και άλλες δόσεις. Εγώ κάνω απόλυτη διάκριση ανάμεσα στις εξωτερικές εξελίξεις και εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα αυτή. Γιατί στην Ουκρανία λένε πολλοί ότι αν δεν καταπολεμηθεί η διαφθορά, αν δεν μειωθεί η δύναμη των ολιγαρχών, δεν θα αλλάξει τίποτα στη χώρα μας. Στην ίδια την Ουκρανία. Ακόμα και το επιτελείο συμβούλων Ο Πίτερ Μπάλας, με τον οποίο συμμετέχει στο monitoring group, με αυτόν συζητήσαμε και είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ήλπιζα να μπορέσω να συνδιαλεχθώ μαζί του για την προετοιμασία της σημερινής συζητήσεως. Δεν πρόλαβα, αλλά ελπίζω να το κάνω τις επόμενες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, ως τροπολογία, εγώ θέλω μια συγκεκριμένη μνήα των όρων και προϋποθέσεων υπό τους οποίους χορηγείται η μακροοικονομική στήριξη. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Ο κύριος Ζατό προβλεπόταν εκ μέρους των Πρασίνων. Α, εσείς κύριε. Κλάους Μπούχνερ λέγομαι κυρία Πρόεδρε. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχύτητα της δράσεώς της. Μία ερώτηση μόνο. Πρόκειται και πάλι για δάνεια. Η Ουκρανία είναι σε κάποιο προβλέψιμο βάθος χρόνου σε θέση να επιστρέψει τα δανεικά ή μήπως την φέρουμε σε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στην Ουκρανία με τον δανεισμό αυτό. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να μπει εδώ και για την επιστροφή των δανεικών. Κατά τα άλλα, εμείς οι πράσινοι συμφωνούμε με την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Η πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν άλλο για την ομάδα δηλαδή EFDD. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάκελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι πιο πολλοί τα είπαν όλα. Συμφωνώ με το κατεπήγον, αλλά μην λησμονήσουμε μια άλλη κατεπίγουσα υπόσχεση που δώσαμε, ότι η πολιτική γειτονία μας θα διαμορφωθεί με πιο συγκεκριμένες αρχές. Πώς θα γίνει αυτό στο πλαίσιο της βοήθειας προς την Ουκρανία, για να διαθέσουμε κάποιους από τους πόρους αυτούς έτσι ώστε να στηριχτούν μεταρρυθμίσεις κράτους δικαίου, ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ. Άλλη ερώτηση είναι ότι στην συμφωνία Μίνσκ, που είναι σημαντική βέβαια, για εκεχηρίες, πολιτικές λύσεις κλπ. Υπάρχουν και κάποια λόγια μέσα εκεί για την εμπορική συμφωνία που έχουμε με την Ουκρανία και που με ανησυχούν, διότι περιλαμβάνονται κάποιες παρατηρήσει που λένε ότι θα διεξαχθούν συζητήσεις με Ρωσία και Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίε που ενδέχεται να προβάλλει η Ρωσία. Ίσως βέβαια να μην είναι η σωστή στιγμή τώρα για να πούμε σε λεπτομέρειες της συμφωνίας Μίνσκ, αλλά προσοχή συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε, να επαγρυπνούμε και να μην τροποποιήσουμε τις περιστάσεις σχετικά με την προτιμησιακή συμφωνία για ένα μισή χρόνο που έχουν αφαιρεθεί τώρα από τη συμφωνία αυτή. Και ίσως σε ιστερότερο στάδιο να πρέπει να επανέλθουμε να δούμε τι συμβαίνει επί της λεπτομέρειας. Ευχαριστώ. Πρέπει να δώσω το λόγο στον εισηγητή, η Κομισιόν, στην οποία αφαιρέθηκαν διάφορες συνάδελφοι. Ε, thank you, ε, Mr. Chairman. Just, ε, ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα, μεθοδή ελέγχου που υλοποιεί η Κομισιόν στο 2-2 της πρότασης. Βεβαίως εδώ έχουμε διάφορες διατάξεις σχετικά. Να πω λοιπόν καταρχάς ότι ακόμα και πριν από αυτή την επιχείρηση και την υιοθέτησή της η Κομισιόν έκανε μια λεπτομερή αξιολόγηση των κυκλωμάτων διεθνών συγγνώμη, ιδιωτικών και δημοσίων διαδικασιών διαχείρισης. Αξιολογήσαμε, αλλά θεωρήσαμε ότι ο κίνδυνος είναι λογικός. Και είπαμε προηγουμένως στις προτεραιότητες μας είναι η ενίσχυση του κυκλώματος διαχείρισης, δημόσιας διαχείρισης μέσω εσωτερικών ελέγχων, εξωτερικών ελέγχων, οικονομικού ελέγχου κλπ. Το ίδιο και το ΔΝΤ του και η Παγκόσμια Τράπεζα. Βεβαίω για τι εγγύησει για την χρήση των κονδυλίων αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο φορολογικό πλαίσιο που συσχετίζεται βεβαίω με αυτό που κάνει και λέει το ΕΜΕΦ, δηλαδή η λιτότητα, σωστή χρήση των κονδυλίων κλπ. Επίσης, να σας πω ότι το ελεκτικό συνέδριο επιβλέπει την λειτουργία αυτών των μακροοικονομικών επιχειρήσεων και βεβαίως κάνει εις βάθος ελέγχους και ελέγχους αποτελεσματικότητας που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα τη συνδρομή μα ευρύτερα δηλαδή πέραν της μακρονομικής αλλά μακροοικονομική και λόγω της σημασία της αποτιμάται και η επίπτωσή της σε τομείς όπως ε, το ενέργειας, διαχείριση των δημοσίων οικονομικών κτλ. Οπότε έχουμε σημαντικές εγγύησεις. Βεβαίως σε περίπτωση όπου διατυπώσουμε παρατυπίες τότε ο ρόλος της Όλαφ είναι καταλητικός. Αυτός απάντησε στο ερώτημά σας. Επίσης είχαμε μια ερώτηση από τους πράσινους για τους κινδύνους σε σχέση με το δεχόμενο με πληρωμή των δανείων. Όπως περιέγραψα προηγουμένως, η χώρα βρίσκεται ε, υπό σοβαρή σοβαρότατη οξία κρίση. Παρ' όλα αυτά, τα επίπεδα χρέους αυξάνονται αλλά όχι τόσο όσο σε άλλες χώρες με αντίστοιχες ε, κρίσεις. Έχουμε και κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου και κυρίως η ύπαρξη προγράμματος το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί με πιο μακρόπνοη προοπτική, βεβαίω θα μειώσει και τους κινδύνους μια αποπληρωμής. Ξέρετε επίσης ότι γίνεται και μια συζήτηση για πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά έχουν γίνει μόνο συζητήσεις γι' αυτό μέχρι τώρα. Και αυτό ενδεχομένω θα μπορούσε να επηρεάσει και την αποπληρωμή του δανείου των τριών δις προς την Ουκρανία. Αλλά δεν προγραμματίζουμε κάποια αναδιάρθρωση της πληρωμής αυτή τη στιγμή, γιατί το δάνειο αυτό έχει δοθεί υπό μορφή ομολόγων κτλ. Δεν ε, προβλέπουμε πάντως την ύπαρξη προβλημάτων σχετικά. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά ε, καλύπτονται και από το Ταμείο Γεήσεων το οποίο βεβαίως ε, περιορίζει και την δυνατότητά μας να δημιουργήσουμε χρέος μέσω των παροχών μας στην Ουκρανία. Γιατί ακολουθούμε ένα ποσοστό 9% έκθεση εκείνη τη χώρα. Υπάρχουν βέβαια κίνδυνοι, όμως η κατάσταση είναι δραματική και θεωρείται πολιτικής προτεραιότητας αυτή η αρρώγη. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένω μπορεί να αποφασίσει πολιτικά να αυξήσει κάπω την έκθεση κινδύνου. Αλλά όσον αφορά το μακροοικονομικό πλαίσιο και το δούνου του που σύμφωνα με την, με την αποτίμησή του η μείωση του χρέου είναι εφικτή σε λογικό χρονικό διάστημα στο 70% και αυτό νομίζω μείνει το κίνδυνο. Τέλος, σχετικά με την Συμφωνία Μίνσκ να πω ότι βεβαίως στην πολιτική της Κομισιόν της Ένωσης δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της ε, συμφωνίας προσχώρησης. Τώρα, οι ανησυχίες της Ρωσίας βεβαίως θα ληφθούν υπόψη υπό την ευελιξία που παρέχει η τωρινή συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης βεβαίως. Δεν θα ήθελα όμως να πάω εδώ σε λεπτομέρειες για αυτή την απόφαση γιατί αφορά περισσότερο τους συναδελφούς συμπεριγνώμονες για το εμπόριο. Για τις αρχές, για θέματα αρχών τώρα, το πώς σχετίζονται όλα αυτά με το MFA. Εσείς επικεντρώνεστε περισσότερο στις πολιτικές πτυχές και όπως είπα προηγουμένως αυτή η επιχείρηση δεν θα έχει προταθεί ποτέ χωρίς να έχει προηγηθεί η διαβούλευση με την υπηρεσία εξωτερική δράσης ώστε να τηρηθούν οι απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις. Η υπηρεσία αυτή εμπλέκεται σε όλη τη διαδικασία, σε όλα τα βήματά της. Πριν υπογραφεί το μνημόνιο, πριν γίνει οτιδήποτε, θα υπάρξει διαβούλευση με την υπηρεσία εξωτερική δράση και με τους νομοθέτες. Και αυτό νομίζω παρέχει εγγύησει ώστε η επιχείρηση αυτή θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές μας όσον αφορά και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που όπως γνωρίζετε θα αποστηρίξουμε και θα ενισχύσουμε την πρόοδο μέσω της οικονομικής αυτής ατζέντα και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι και εμείς αλλά και η κοινωνία να προχωρήσουμε αυτή την οικονομική ατζέντα και τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν καταρχάς για τη δουλειά που έκανε για την προετοιμασία και τη δεκμήρωση αυτού του φακέλου. Να ευχαριστήσω και τους κοιόδης που αποδέχονται έτσι αυτή, την κοινή μας άποψη. Είναι πολύ σημαντικό για την Ουκρανία να υπάρχει ομοφωνία στις θέσεις μας. Και αυτό είναι το κύριο μήνυμα που στέλνουμε. Συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Για τις επιμέρους ερωτήσεις και ζητήματα, θέματα ελέγχου, αν η κατάσταση δεν ήταν τόσο τρομακτική, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση πιο εύκολα για τον έλεγχο, διαφορές προσεγγίσεις ε, για τον έλεγχο των δαπανών, τι πάει σε ιδιωτικές ε, τσέπες κτλ. Όμως μιλάμε τώρα για την επιβίωση της χώρας και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν είναι καταλληλότερη στιγμή να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και νομίζω συμφωνείτε όλοι. Θα συμφωνήσω λοιπόν με αυτή τη συζήτηση όταν η κατάσταση σταθεροποιηθεί και όταν θα συζητήσουμε και θα μιλάμε για το πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Τώρα όμως μιλάμε για το πώς θα τη σταθεροποιήσουμε επειδή έχουμε ένα κατήφορο. Συμφωνία Μίνσκ τώρα. Ίσως βρίσκεται εκτός παρόντος πλαισίου αλλά έχω μεγάλες εμφωλίες κατά πόσο η συμφωνία του Μίνσκ θα προχωρήσει γιατί και η κατάπαυση του πυρός αφισβητείται και δεν ξέρω κατά πόσο καν θα καταλήξουμε σε συζήτηση για την εξέταση της συμφωνίας σύνδεσης ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις ανησυχίε της Ρωσίας. Αλλά νομίζω τα πιο σημαντικά ζητήματα από αυτά αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Λασπέργης. Θα κλείσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 25 του Φλεβάρι το μεσημέρι συζήτηση και ψηφορία 18-19 Μαρτίου στην Επιτροπή και Ολομέλεια, δεύτερη Ολομέλεια Μαρτίου, 1η Απριλίου. Σας ευχαριστώ όλους. Προτείνω τώρα αγαπητοί συνάδελφοι να περάσουμε στο σημείο 6 της ημέρης διαταξής, δηλαδή η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Έκθεση πρωτοβουλίας της, της Επιτροπής Ήτρε μετά από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμεί προσθέτουμε εδώ την διάσταση του εξωτερικού εμπορίου σε μια, στα πλαίσια μιας σφαιρική πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια. Σόλτ είναι ο κύριος εισηγητή και θα δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Merci, Madame euh, Chair. Πρώτα ευχαριστώ. Dear colleagues, we are discussing today our draft Συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα την έκθεση Ιδέας πρωτοβουλία για την Ενέργεια ανταποκρινόμενη στην ανακοίνωση τη Κομισιόν του Μάη πέρσι αλλά και τι παραμονέ τη συζήτηση για θέματα ενεργεία στην Ένωση. Να το τονίσω αυτό επειδή θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνουμε πολύ γρήγορα με τις συζητήσεις και τα συμπεράσματά μας για την ασφάλεια, την ενεργειακή, χωρίς να γνωρίσουμε λεπτομερώς τις προτάσεις οι οποίες θα προέλθουν από την Κομισιόν αυτή ή την επόμενη εβδομάδα. Ήδη είχαμε μια συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών και έχουμε τις συμβολές τους ήδη στο πρώτο σχέδιο του κειμένου. Αλλά πρέπει να πάμε γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Πάντως είχαμε ένα περιορισμό 500 ε, χαρακτήρων για αυτή την πρόταση και αυτό με υποχρεώνει να επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα ζητήματα γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να περάσουμε αυτή τη γραμμή. Οι σκιώδεις επίσης έλαβαν και δικές μου προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν ως Θα πρέπει ως Επιτροπή να εστιάσουμε στα θέματα που αφορούν το εμπόριο. Θα δείτε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπογραμμίζω το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας ως θέμα παγκόσμια σημασίας και για την Όση και για τους εταίρους της και για την ανάγκη σύναψης εταιρικών ενεργειακών σχέσεων. Η πρόσβαση στην ενέργεια ως ανθρώπινο δικαίωμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, εξοικονόμηση ενέργειας ως τρόπος μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές και τη μείωση του εμπορικού συζυγίου των χωρομελών. και τέλος νέα μορφή ενέργειας σε σχέση με τις τεχνολογίες και ως ευκαιρία εξαγωγών από την Ένωση και σε συνεργασία με τρίτους. Αγαπητοί συνάλφοι, η ενέργεια αυτή τη στιγμή συζητείται ευρέως ως θέμα πολέμου και ειρήνης. μετά από αυτά που είπαμε κιόλας για την Ουκρανία. Η στρατηγική ασφάλεια ενέργεια έχει στόχο το 2030 και κατά την άποψή μου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας πέραν των τωρινών κρίσεων και να υπογραμμίσουμε το ότι οι εμπορικές μας συμφωνίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ένα μέλλον βιώσιμο για την ενέργεια και την βιώσιμη κατανόηση της ενεργειακής, ε, του ενεργειακού εφηβοδιαωσμού. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για περιπτώσεις συνεργασία σε αυτή την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Θα δώσω το λόγο για το έλξο στον κύριο Φέρνελ που αντικαθιστά τον κύριο Σάνφελντ. Ευχαριστώ. Είμαι ο κύριος Σάνφελντ. Έτσι να με κλάβετε. Καταρχάς, ο θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη επειδή δεν μπορεί να συμμετάσχει σήμερα, αλλά ω σκιώδη θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Σόλτ, τον εισηγητή για την δουλειά του. Καλωσορίζει το γεγονό ότι η γνωμοδότηση υπογραμμίζει τον κύριο ρόλο του εμπορίου στην ενεργειακή ασφάλεια τη Ένωσης. Έχουμε ολόκληρα κεφάλαια ενέργεια στι συμπορικές Φωνη που συνάπτει η Ένωση η ανάγκη ύπαρξη ενεργειακή αγορά μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επίση και να περιληφθεί στι ε, διαπραγματεύσει. Είναι η απόψη του. Επίση, θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα και διατάξει που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση και είναι καταρχά η εστίαση στι ΑΠΕ, στην ίδια τη στρατηγική αλλά και στα πλαίσια τη νομοδότηση. Βεβαίω, ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν αφορούν το όφελος των ΑΠΕ. Υπάρχουν πολλά, διορθώνει μιλήτες, υπάρχουν πολλά ωφέλη από τι ΑΠΕ. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει όμω να προσεγγιστούν από ιδεολογική σκοπιά. Όταν συζητάμε για την ενεργειακή ασφαλεία στην Ένωση, να μην ξεχνάμε και τον ρόλο των ντόπιων ορυκτών καυσίμων λόγω του χαμηλού κόστου εξόρυξη και μεταφορά και αποθήκευση. Αν αποφασίσουμε να περιοριστούμε, να περιορίσουμε τον ρόλο των ντόπιων ρηκτών καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως στο μέλλον αυτό σημαίνει ότι θα εξαρτώμαστε πλήρως από τις αγωγές που έχουν βεβαίω αρνητικό αντίκτυπο στην ενεργειακή μας ασφάλεια. Ένα άλλο σημείο ο κ. Παντικαθιστό θεωρεί ότι είναι σημαντικό θα πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι θα πρέπει να απαλληφθεί η ενεργειακή, ασφάλεια, φτώχεια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αναφέρεται το σχέδιο γνωμοδότησης, παρόλα αυτά ο στόχο αυτό θα πρέπει να βασίζεται και στην πραγματικότητα. Γι' αυτό ακριβώ είναι απαραίτητο να φτιάξουμε την πολιτική στην Ένωση για τα ενεργικά θέματα χωρί να μειώσουμε την οικονομική ανταγωνιστικότητα τη Ένωση παγκοσμίω. Κατά το οποίο θα οδηγούσε στην αύξηση τη ε, και τη στόχη, συμπληρωμένη και τη ενεργικής στόχη των πολιτών. Γι' αυτό ακριβώ θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι θα θέλαμε να καταθέσουμε περαιτέρω τροπολογία στη συνέχεια. Και θα επανέλθω και εγώ σε αυτό το θέμα αργότερα. Ναι. Ε, θα έρθει και η σειρά σου μετά από τους κοιόδες. Δαβίδ Μαρτίν, που αντικαθιστά τον κύριο Λάγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μετά, εξ ονοματός του, του ιδίου, θα λάβει και αυτό το λόγο. Να ξεκινήσω καταρχάς εξ του Μπέρντ να ευχαριστήσω κύριο Σόλτς για την καλή συνεργασία. Χαίρετε ο συνάδελφος για την συμφωνία αυτή, για την γνωμοδότηση μάλλον και το κείμενο που συνέταξε ο Συγητή, ώστε να συνεργαστούμε ως Ένωση σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς προκλήσεις στο πεδίο της ενέργειας, στην καταπολέμηση της ενεργειακής ε, φτώχειας παγκοσμίω. Χαίρεται ιδιαίτερα για το γεγονό ότι το σχέδιο γνωμοδότηση αναφέρεται ιδιαίτερα στην ενεργειακή απόδοση και στι ΑΠΕ, στο σημείο 6 του κειμένου. Και κατά την του, η εξοικονόμηση ενέργεια είναι η καλύτερη λύση και η ενεργειακή απόδοση είναι ο καλύτερο τρόπο για να ασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια. Η εξοικονόμηση όχι μόνο μα βοηθάει στο να πετύχουμε του στόχου του περιβαλλοντικού, αλλά μα επιτρέπει επίση να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ανάπτυξη και στην καινοτομία του τομέα τη ενέργεια και τη ενεργειακή απόδοση, ε, βοηθώντα να διασφαλίσουμε και να πετύχουμε την ε, τεχνολογική έτσι, πρωτοπορία τη ένωση σε αυτά τα θέματα. Επίση, με χαρά βλέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο γνωμοδότηση το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεργασία ε, στον τομέα και στο πεδίο της διοργανικής διεθνούς συνεργασίας ώστε να υπάρχει διαφάνεια και θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως ισχυρή νομοθεσία όπως επίσης και σωστή εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό το σημείο θα καταθέσει μια επί τροπολογία. Τελευταίο του σχόλιο είναι το ότι οι εμπορικέ συμφωνίε θα πρέπει όλε να περιλαμβάνουν μελλοντικά κεφάλαια ενεργειακά ώστε να διαφοροποιηθούν ενεργειακέ πηγέ, να διασφαλιστούν προδιαφέ ποιότητα για την ενέργεια και να είναι βιώσιμη η παραγωγή ε, ενέργεια και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα καταδεχθεί και επί του, του τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζαρατήλουσερ, ο οποίο θα μιλήσει εξωματό του του ιδίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Σόλτς περιλαμβάνει κάποια σημεία κλειδί. Να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Ένα απολύτως κύριο σημείο είναι το σημείο 3 όπου υπογραμμίζει το ότι το εμπόριο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την βασική ιδέα στις δηλώσει μας, στη στάση μας και στις τροπολογίες μας. Νομίζω ότι το επίκεντρο για μας είναι η ενεργειακή ασφάλεια μαζί με την οικονομική δραστηριότητα και την, και την ανταγωνιστικότητα. Και θα πρέπει να εστιάσουμε στο να διασφαλίσουμε σίγουρη και σταθερή πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει επίσης να αποβλέπουμε στην μείωση της εξάρτησης από ένα και μοναδικό προμηθευτή ή από ένα και μοναδικό σημείο διέλευσης. Επειδή αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστρατήγηση, η κατάχρηση της δεσπόζας αυτής στην αγορά. Θα πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν νέους εταίρους σε άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν το ρόλο προμηθευτών ενέργειας, Αφρική, Ασία κτλ. Και Αμερική βέβαια. Και αυτό θα έπρεπε να περιληφθεί σε κάποιες από τις τροπολογίες μας. Δεύτερον, και πάλι για το ρόλο του εμπορίου θα πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών εμπορίου, των εμπορικών πολιτικών, το οποίο σημαίνει ότι τα νοσιακά και άλλα εργαλεία θα πρέπει να αποβλέπουν στη βελτίωση της πρόσβασης για την Ένωση στην αγορά, κάτι το οποίο παίζει τρολό βράχη μέσω πρόθεσμα. Τρίτον, οι διεθνείς κανονισμοί. Γιατί σε πολυμερό επίπεδο δεν ρυθμίζεται η ενέργεια. Οπότε θα πρέπει να γίνεται αυτό με τρόπο σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διεθνές πλαίσιο κανόνων που θα αφορούν τις τεχνολογίες ενέργειας, τα προϊόντα ενέργειας και βεβαίως αυτό ιδανικό θα ήταν να προέρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ώστε το πλαίσιο αυτό να συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας, της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας και στη μείωση των εντάσσεων μεταξύ των χωρών μελών εντάσσεων που απορρέουν από το εμπόριο ενέργειας, θέμα που θίγει ο κ. Σότς στην νομοδότησή του στο σημείο 5 και στο 6. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτής Αυτές οι τρεις κυρίως πτυχές θα πρέπει να ενισχυθούν στην γνωμοδότηση και αυτό ακριβώς θα πρέπει να ακολουθήσουν αντιστοιχέ τροπολογίες τις οποίες θα τις καταθέσουμε αντιστοίχως ώστε να έχουν έτσι και την δέουσα υποστήριξη από την Επιτροπή μας και να γίνουν αποδεκτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ολιαράν για το Αλντέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σόλτς για το σχέδιο και την ταμάση συνεργασία που είχαμε. Τρία σημεία για αυτό το σχέδιο. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι αρκετά ισορροπημένο και συνδυάζει θέματα τα οποία είναι σημαντικά για το διεθνές εμπόριο. Ένα από αυτά βεβαίω είναι το ότι η Ευρώπη σήμερα εξαρτάται υπερβολικά από τα ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα έπρεπε να έχουμε ενεργειακά κεφάλαια στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών όπου εμπλέκεται η Ένωση. Το τύπο, ας πούμε με την αύξηση ενεργειακού εμπορίου και εμπορίου πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλάβει αυτό το σημείο. Δεύτερον, για το 6 από τις προτάσεις του κ. Σόλτς συμφωνώ παρόλο που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο ως σημείο και μακρόπνο να μην μιλήσουμε για ΑΠΕ και απόδοση παγκοσμίω είναι σημαντικό να τεθεί και στο πλαίσιο της Ευρώπης. Πρώτα να αναφέρει το σημείο 1. Και τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι βεβαίως χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες ενεργειακές πολιτικές όμως καμιά φορά οι δράσεις της Ένωσης είναι κάπως δίσκαμπτες και όχι πάντοτε συνεπείς με τους στόχους των πολιτικών μας. Και εδώ, καθώς κοίταζα το σχέδιο της Ίντρε, νομίζω θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο της ΑΠΕ και ο κύριος Γιούνκερ νομίζω έκανε μια έκκληση είτε θα γίνει η Ένωση ο υπαριθμό ένα παραγός ΑΠΕ είτε όχι. Κατά την απόψή μου το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να περιλάβει αυτή την αναφορά στις εκθέσεις και στα ψηφίσματά μας. Γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι που ο κ. Σόλτ στο έγγραφό του το υπογραμμίζει αυτό το σημείο περισσότερο από το έγγραφο της ΣΥΝΤΕ. Περιλαμβάνοντας βεβαίως και την καθαρή ενέργεια και την ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον, κάτι το οποίο αναφέρεται στο σημείο 7 του κείμενου του κ. Σόλτ. Και ένα τελευταίο σημείο γενικότερο. Για το έγγραφο της ΙΝΤΕ γίνεται συζήτηση για μια ένωση ενεργειακής, ενεργειακών επενδύσεων. Γιατί να μην προβλέψουμε μια συζήτηση με μεγαλύτερο ρόλο της Ένωσης. Έχουμε μια Ένωση κεφαλαίων. Έχουμε τραπεζική Ένωση. Επενδυτική Ένωση γιατί να μην κάνουμε και μια ένωση επενδύσεων ενεργειακών ώστε να, αποτελε... να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για, για τους πάσους ο κύριος Μπούχνερ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας έκθεση. every single point of it, but ε, ε, πρέπει να σας πω πως έχουμε κάποια θέματα τα οποία θέλουμε να ξεκαθαρίζονται περισσότερο και αυτή είναι η άποψη ε, των σοσιαλδημοκρατών. Καταρχήν η ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζεται στην αποδοτικότητα, στη ΣΑΠΕ και στην διασυνδεσιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων έτσι ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από αυτού του είδους συνεργειακούς πόρους. Επίσης, μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Και αυτό είναι ένας στόχος μέσω της αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας. Έτσι ώστε να μην εξαρτώμεθα τόσο από τις εισαγωγές καυσίμων. Η σύναψη συμφωνιών, εμπορικών συμφωνιών με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να συνάδει με τις εσωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια, κάποιες μέθοδοι ε, εξόρυξης που δεν μπορούν να γίνουν ε, ποδεκτές. Για παράδειγμα, ε, συστολιθικό αέριο. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην εξόρυξη, στην περίπτωση εξόριξης ουρανίου για μία και μοναδική εγκατάσταση, για ένα και μοναδικό σταθμό ε, πυρηνικής ενέργειας χρειάζεται να εξοριχθούν κατ' έτος 500 εκατομμύρια τόνοι ραδιενέργειας υλικό με τεράστιες επιπτώσεις για το περιβάλλον αλλά και για τους ε, κατοίκους της γύρω περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν στις ε, εμπορικές συναλλαγές που έχουμε με τις χώρες αυτές για τα υλικά αυτά να ισχύουν ίδιοι οι κανόνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την εμπορική μας πολιτική λοιπόν έτσι ώστε να καλύπτει το στόχο της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να πω πως η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ελεύθερη εκπομπών διοξιδίου και αν λάβουμε υπόψη όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας από την εξόριξη τήξη ουρανίου, εμπλουτισμό, κατασκευή σταθμών κτλ. θα καταλήξουμε στο 32 με 60 γραμμάρια διοξιδίου ανά κιλοβατόρα. Τα νούμερα αυτά εξαρτώνται βεβαίως και από το είδος ουρανίου που εξορίσετε και από την ε, τύπο εμπλουτισμού που επιλέγετε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις άλλες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αν αυτό είναι συγκρίσιμο με τις εκπομπές ε, διοξιδίου εκεί. Έχουμε δηλαδή εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο που παράγουν μόνο ηλεκτρισμό, όπου εκεί οι εκπομπές είναι υψηλότερες. Και ε, εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερού που παράγουν και θερμότητα, ναι, δηλαδή θερμοηλεκτρική σταθμή με καλύτερες επιδόσεις. Δεν συζητώ βέβαια τις πολύ καλύτερες επιδόσεις των αιωλικών πάρκων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα συγκεκριμένα νούμερα πριν αποφασίσουμε. Το επόμενο σημείο είναι τι θα γίνει και πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ενέργειας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως τουλάχιστον σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, με, χωρί, χωρίς μάλλον εξωτερική βοήθεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που χρειαζόμαστε για ε, ένα συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων. Άρα λοιπόν αυτό που λείπει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ε, γίνει η αιωλική ενέργεια αέριο ε, και μετά ε, ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία είναι πολύ γνωστή και το μόνο που χρειάζεται έτσι ώστε να εισαχθεί στην παραγωγή είναι να είναι παράλληλα και κερδοφόρα. Και αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται λόγω κάποιας ε, πολύ περίεργης νομοθεσίας που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους μεταβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την πυρηνική ενέργεια, εκεί θα πρέπει η παραγωγή να ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες του ΠΟΕ, δηλαδή σε επίπεδο ε, επιδοτήσεων, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε μια πιο διευρυμένη προσέγγιση. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι οι επιδοτήσεις για όλα, όλες τις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί εδώ τα νούμερα είναι ιδιαίτερα υψηλά και θα το έχετε καταλάβει αυτό από τη συζήτηση που έγιναν τον περασμένο μήνα. Eight times as much Έχουμε λοιπόν για παράδειγμα τιμές feed-in στο δίκτυο που είναι 8 φορές υψηλότερες από αυτές για την αιωλική ενέργεια. Άρα λοιπόν οι επιδοτήσεις και τέλος το κόστος αυτών των ε, διαφορετικών μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ευθυγραμματίζεται με τους κανόνες του ΠΟΕ. Merci, ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Σόλτς για τη δουλειά και την διάθεση που έδειξε. Οι αμφιβολίες μου είναι κυρίως δύο για αυτό το θέμα, όπως είπα στην προηγούμενη συνάντησή μας των σκιωδών. Καταρχάς, τοπικοί πληθυσμοί. Νομίζω ότι σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθησαν εμπλέκοντας στα ενεργειακά τους ντόπιου πληθυσμού. Πετύχαμε πολλά με την ενημερώση των πολιτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξοικονόμηση και καλύτερη χρήση της ενέργειας. Όταν μιλάμε όμως μετά για εμπόριο ενέργειας στην Ευρώπη και εκτός, ξεχνάμε τελείως τους ντόπιου. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις υποδομές. Νομίζω εκεί δεν γίνεται να μην συμμετέχουν οι πολίτες και να υπάρχει δυνατότητα από κάτω να υπάρχουν προτάσεις ιδιαίτερα όταν αυτέ οι υποδομές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους ντόπιου πληθυσμούς. Η δεύτερη μου αμφιβολία αφορά ένα ζήτημα που σχετίζεται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Μιλάμε πολύ για υποδομές, συζητάμε πολύ το ρόλο τους, ξεχνάμε όμως ότι η ενέργεια εξαρτάται και από την έρευνα αν δεν επενδύσουμε εκεί δεν θα βγούμε από δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό είναι κάπως αντίθετο με τις επιλογές της Κομισιόν, ιδιαίτερα με το σχέδιο Juncker που κάνει περικοπές στον τομέα αυτό. Περικοπές όσον αφορά τις διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Το υπενθυμίζει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, υπογραμμίζοντας ακριβώς αυτή την πτυχή. Νομίζω ότι σε μια τέτοια έκθεση δεν μπορούν να λείπουν αυτά δύο σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι λοιπόν έχουν το λόγο. Θα προσπαθήσω να εστιάσω στα θέματα εμπορικής πολιτικής σε σχέση με την εξασφάλιση του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Νομίζω πως το σχέδιο του κειμένου είναι εξαιρετικό και θα ήθελα να συνταχθώ με μία άποψη την οποία σας διάβασα προηγουμένως παρόλο που δεν ήταν δική μου. Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην αντιμετώπιση του θέματος και τις εμπορικές ε, συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα με τη ΣΥΠΑ, μήπως και εκεί μπορούμε να εντάξουμε και ένα ενεργειακό κεφάλαιο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για ασφάλεια, ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε καταρχήν τις διάφορες τα, ταρίφες που έχουμε στην ενέργεια. Ε, εκεί δεν ισχύουν ποσοστώσεις γιατί θέλουμε ευθυνές εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πρέπει να σας πω ότι για την πράσινη τεχνολογία εκεί ισχύουν κάποιοι περιορισμοί στα μέτρα και στις τιμές λόγω ε, προσπαθειών που γίνονται ε, για dumping και είναι κάποια ανταλλακτικά για ε, ανεμογεννήτριες, είναι ε, κάποια φωτοβολταϊκά πάνελ κτλ. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση. Διαπιστώνω πως για παράδειγμα για το μαγνητικό χάλιβα που είναι από τα πιο σημαντικά ανταλλακτικά που χρειάζεται όταν κανείς προσπαθεί να μεταφέρει ενέργεια ε, στα πλαίσια δικτύων ε, πρόκειται να, δικαστεί μια, να ακουστεί μάλλον μια υπόθεση ε, anti-dumping. Οπότε ας δούμε πού βρίσκεται το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπου σας είπα ότι ενδεχομένως να υπάρξει και τέτοια υπόθεση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τεράστιες επενδύσεις πάντως για να είμαστε ενεργειακά ασφαλείς. Πράσινη τεχνολογία, ε, υποδομές, δικτύων και παράλληλα υπάρχει πολύ μεγάλος πολιτικός κίνδυνος και πολιτική αβεβαιότητα γιατί εμείς είμαστε πολιτικοί και δεν συμφωνώ με καμία από τις ε, παρατηρήσεις που έκανες εδώ στη δεύτερη παράγραφο που λες πρέπει να ενισχύσουμε τον πολιτικό έλεγχο και την πολιτική ρύθμιση. Θα έλεγα όχι, η ενεργειακή παραγωγή είναι ένας κλάδος που ρυθμίζεται πολύ αυστηρά σε σχέση με τους υπόλοιπους ε, κλάδους στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν το θέμα της προστασίας των επενδύσεων στην Ευρώπη και ειδικά για τις επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία στον ενεργειακό κλάδο ίσως να είναι το πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση για την προστασία των επενδυτών στην συμφωνία μας με τη ΣΥΠΑ. Εάν θέλουμε όμως να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια που υπάρχει μεγάλο πολιτικό, μεγάλος πολιτικός κίνδυνος, ίσως ε, αυτό είναι ένας τρόπος για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε και σε εμά. Και αυτή ήταν και η τελευταία μου παρατήρηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτιν, όχι. Ο κύριος Μπρουτινάρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να παραμείνω στα χωράφια της Ίντα και να μην μπόσφια για ενεργειακά θέματα, γιατί όταν μιλάμε για μια στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, νομίζω ότι σήμερα πιο πολύ από ποτέ η ενέργεια σημαίνει ασφάλεια και δεν θα τα σχολιάσω αυτά. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει μια δραματική ανάγκη να συντονιστούμε σε επίπεδο εξωτερικών ε, πολιτικών, πολιτικών ασφάλειας και πολιτικών διεθνούς εμπορίου έτσι ώστε ο δικός μας ρόλος να γίνει πιο σημαντικός. Το πακέτο για την, Ευρωπαϊκή, για Ενεργειακή Ένωση σύντομα θα εγκριθεί και στα πλαίσια του πακέτου αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει το μελλοντικό της σχεδιασμό για πολλά ενεργειακά θέματα και την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Αυτό το είπε και ο κύριος ε, Γιούνκερ και η κυρία Μογκερίνη και τη δέσμευση αυτή ανέλαβε και η Επίτροπος Μάλστρομ όταν πέρασαν από τις ακροάσεις. Άρα λοιπόν ας παραμείνουμε σε αυτά τα πλαίσια των δεσμεύσεων που ανέλαβαν στην αρχή της θητεία του. Το δεύτερο θέμα είναι να μειώσουμε την βαριά εξάρτηση από ένα μοναδικό προμηθευτή. Δεν θα κατονομάσω αλλά θα πρέπει στο μέλλον να μοιάσουμε αυτή την πραγματική εξάρτηση που έχουμε από ένα και μόνο προμηθευτή. Πώς, βρίσκοντας εναλλακτικέ πηγές, εναλλακτικέ οδούς μέσω της σύντα. Δηλαδή, μέσω της πολιτικής μας για το διεθνές εμπόριο. Όχι να ακούμε αυτά που λέει η Ήτρε, μέσω της δικής μας προσπάθειες για διεθνή εμπορικές σχέσεις και συμφωνίες. Έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας, τις τρίτες χώρες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι διμερός ή σε μικρό μαδούλες ευρωπαϊκών χωρών διαφορετικά θα είμαστε ένα σωματείο χαμένων και καταλαβαίνετε τι τροπή θα λάβουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ημών και της Γκάσπρομ. Αν ως εθελοντές προσφέρουμε αυτούς οι οποίοι λιγότερο είναι διαθεθειμένοι να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία και την Γκάσπρομ. Είναι ουσιαστικό κατά τη γνώμη μου ότι τα ενεργειακά κεφάλαια να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και στην TTIP γιατί έτσι η Ευρώπη θα καταφέρει να μειώσουμε περαιτέρω την εξάρτησή μας, θα προωθήσουμε τις διεθνείς μας εμπορικές πολιτικές στο χώρο της ενέργειας, εμείς θα προτείνουμε και εμείς θα εφαρμόσουμε τους δικούς μας κανόνες έτσι ώστε να καταφέρουμε την ενεργειακή ασφάλεια μέσω των διεθνών συμφωνιών. Ευχαριστώ τον κύριο Σόλτς για την συνεισφορά του και βεβαίω θα καταθέσω επιπλέον τρόπολογίε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρόσωπο της Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής Δύο λόγια μόνο. Όπως είπαν κάποιοι από τους βουλευτές, το έγγραφο για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για την Ενεργειακή Ένωση θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει η διεθνής διάσταση που λαμβάνεται υπόψη και μία από τις παρατηρήσεις που ακούσαμε είναι πολύ σημαντική ε, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε για την δημιουργία της ε, Ενεργειακής Ένωσης. Ψάχνουμε να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ των διαφόρων προτάσεων των επιτροπών σας. Έγινε μια συζήτηση και στην ΙΜΚΟ και θα, στην Ήτρε θα γίνει μια συζήτηση και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να έχουμε ένα κόνσεπτ της ενεργειακής ασφάλειας που είναι να τον πιο διευρυμένο. Δηλαδή εσωτερική αγορά, διεθνής διάσταση, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αυτή η πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα διάφορα σκέλη είναι για εμάς ε, το στοιχείο που θα δώσει επιτυχία, θα στέψει με επιτυχία τις προσπαθίες μας. Θα σας δώσω λοιπόν και περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της πρότασής μας και βεβαίως θα διαβάσουμε πολύ προσεκτικά και όλες τις τροπολογίες που θα καταθέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής έχει και πάλι το λόγο. Uh, I want to thank all colleagues, Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους ε, για, τα σχόλιά τους και σας, κυρία Πρόεδρε γιατί όντως συμφωνώ είναι πάρα πολλές οι πτυχές της ενεργειακής παραγωγής, του ενεργειακού εμπορίου, του ενεργειακού ανεφοδιασμού, ε, να έχουμε φθηνή προσβάσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες αν μιλάμε για την εμπορική διάσταση. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω. Και έχω μία παρατήρηση στην οποία θα ήθελα να απαντήσω. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα του εκδημοκρατισμού της χάραξης πολιτικής. Θα πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν στο μέλλον. Η ενέργεια και οι ενεργειακέ επενδύσεις συνδέονται και με τα συμφέροντα και την ικανότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια ε, προς όφελος των ιδίων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ε, Προσδοκώ λοιπόν με χαρά όλε τι τροπολογίε, γιατί όπω σα είπα από την αρχή θα πρέπει εμεί μαζί συλλογικά να συνεισφέρουμε με τις δικές μας ιδέες έτσι ώστε την έκθεση αυτή να την εμπλωτίσουμε με την συνεισφορά όλων μας και την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία λείπουν, οπότε ελπίζω πως ε, θα καταφέρει το Κοινοβούλιο να συμπληρώσει ε, τα θέματα αυτά ε, με κάποια επιπλέον στοιχεία και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες. 26 Φεβρουαρίου, 4 η ώρα. Τελευταία ευκαιρία να τις καταθέσετε. Θα περάσει ε, από την Επιτροφή 18 και 19 Μαρτίου προς ψηφοφορία και ολομέλεια του Μαΐου για την τελική ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 6. Το 7, με συγχωρείτε, περιορισμοί σε εξαγωγές και μία πρώτη ανάγνωση του κανονισμού για τα βασανιστήρια κτλ. Για αγαθά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για εκτελέσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο κατευθείαν στην εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που φωτίσατε ένα θέμα εξίσου σημαντικό με πιο περιορισμένο πεδίο από ότι άλλα θέματα, τον κανονισμό αυτό κατά των βασανιστήριων. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κατάλογος με τα αγαθαδητής χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ε, κτλ. Η απαγόρευση των βασανιστήριων και της θανατικής ποινής είναι ένα από τα βασικά ε, τις βασικές και θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής μας πολιτικής, άρα λοιπόν θα πρέπει να απηχείται και από την εμπορική μας πολιτική. Οι στόχοι δεν είναι αμφισβητήσιμοι, αλλά υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα που πρέπει να κοιτάξουμε για να είμαστε πιο ευέλικτοι και αποτελεσματικοί και πιο σύγχρονοι. Χαιρετίζω τις δηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου, είναι πολύ φιλόδοξη ε, στο θέμα αυτό, θα προωθήσουν το φάκελο και θα συνεργαστώ μαζί τους για να καταλήξουμε σε ένα θετικό συμπέρασμα. Η σχετική νομοθεσία αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχουμε μονομερώς εφαρμόσει και είναι διαφορετικό από, τους, από τα καθεστώτα ε, εξαγωγικού ελέγχου των αγαθών διητής χρήσης. Όμως είναι μηχανισμοί που είναι συμβατοί μεταξύ τους, είναι ευέλικτοι και μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις τεχνολογικές εξελίξεις ή τις αλλαγές που βλέπουμε επί τόπου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως δεν θα, υπερβαρύ, δεν θα βαρύνουμε υπερβολικά τις επιχειρήσεις που εξάγουν στον κόσμο και θα πρέπει να ενισχύσουμε την νομοθεσία έτσι ώστε να συνεισφέρει στους στόχους εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει όντως πως χρειάζεται πιο αποτελεσματικός έλεγχος για παράδειγμα, οι εξαγωγές χημικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις θανατηφόρους ε, ενέσεις, αλλά παράλληλα έχουν και νόμιμη χρήση. Ορισμός ε, βασανιστήριων ε, και οποιασδήποτε αναξεπρεπούς μεταχείριση ανθρώπων είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζομαι στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οποιαδήποτε προσφορά δική σας είναι καλοδεχούμενη. Επίσης διαμεσολάβηση και τεχνική βοήθεια για τα προϊόντα αυτά είναι ένας χώρος που θα πρέπει να καλύψουμε ακόμα και όταν δεν προέρχονται τα προϊόντα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει κάποιες υποβοηθητικές εργασίες, χρηματοπιστωτικές, ασφάλεια, διαφήμιση, μεταφορές, προώθηση των προϊόντων αυτών να απαγορευτούν επίσης για να έχουμε ένα σύστημα συνεπές το οποίο θα προσφέρει ίδιους κανόνες σε όλους θα πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία, συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη χορηγούν ή απορρίπτουν αιτήσει για εξαγωγικές άδειες έτσι ώστε να υπάρχει ένας κανόνας που θα ισχύει για όλους. Για τα συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να αξιολογηθούν σωστά αυτά τα προϊόντα, ε, θα πρέπει να αποτανθούμε ε, στη συντεταγμένη κοινωνία, στους εμπειρογνώμονες, ε, στις τεχνικές αρχές, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με μια εξωστραφή φορά για να καλύψουμε και όλες τις πτυχές των ζητημάτων αυτών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο. Δηλαδή, μία επίγουσα διαδικασία θα πρέπει να προβλέπεται. Επίσης, εποπτεία από εμάς και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή για τις αγαθά διτής χρήσης και θα πρέπει οι εξαγωγικές άδειες και οι περιορισμοί σε αυτές να μπορούν να τροποποιηθούν γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που μεταλλάσσεται και είναι εξίσου σημαντικό αυτό όπως και στον κανονισμό για τα αγαθά διτής χρήσης. Και νομίζω ότι υπάρχει μια επικάλυψη μεταξύ των δύο αυτών χώρων και όπου έχουμε αποδείξεις παραβίασης με επιτρεπόμενα υλικά, για παράδειγμα δακρυγόνα που παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν να, για ρήψεις από κοντά, άρα χρησιμοποιούνται πλέον ως όπλο, θα πρέπει να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια για να είναι αποτελεσματική νομοθεσία. Κλείνοντας να σας πω πως οι μηχανισμοί ε, ελέγχου των εξαγωγών για αγαθά που χρησιμοποιούνται στα βασανιστήρια είναι σημαντικοί. Είναι καταρχήν πολιτικής φύσης η συζήτηση και υπάρχει και το θέμα της ε, ε, ε καταδίκης, ε, των απάνθρωπων ε, βασανιστήριων, και η προσπάθεια που κάνουμε του περιορισμού της εμπορίας αυτών των αγαθών είναι ένα μόνο βήμα αλλά πολύ σημαντικό στα πλαίσια ε, των προσπαθειών που κάνουμε ε, ιδιαίτερα στο χώρο αυτό. Merci. Je donne la parole... Daniel Κασπάρη, ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να έρθω σε μια λεπτομέρεια. Η εργασία που μας έχει υποβληθεί είναι καλή. Να δούμε μόνο, να εξασφαλίσουμε δηλαδή, αφενός βεβαίως αποτελεσματικούς εξαγωγικούς ελέγχους και μάλιστα να απαγορεύονται τελείως οι εξαγωγέ σε ορισμένες χώρες, να φροντίσουμε όμως να μην βάλουμε στο ίδιο καλάθι όλα τα προϊόντα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ορισμένα. Παράδειγμα, μπορώ να φανταστώ διάφορα ιατρικά προϊόντα, φάρμακα που η συνήθι χρήση τους είναι ορθή, λογική, καλή, αλλά μπορεί ορισμένοι να τα χρησιμοποιήσουν, να τα καταχραστούν τέλο πάντων για βάρβαρους σκοπούς. Εδώ χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε μια ευφυή λύση, ώστε να μην επιβάλλουμε ρυθμίσεις σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους κατασκευαστές που αφενός δεν πρόκειται λύσουν το πρόβλημα, αφετέρους θα προκαλέσουν μεγάλη, πολύ μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Αν συμφωνήσει καταρχήν η συγγήτρια θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πάντως για τη θαυμάσια έως τώρα συνεργασία. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, David Martin η κυρία Ροντρίγκε την οποία εκπροσωπώ, είναι και ο η εισηγητρία θα συνεργαστεί με την εισηγήτρια. Χαίρεται για αυτή την νομοθεσία κατά των βασανιστήριων. Δύο βασικά σχόλια. Όπως ερμηνεύουμε εμείς τον κανονισμό, επιτρέπει σε μη ευρωπαϊκές εταιρείε να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να διευκρινιστεί εάν θα υπάρξουν και σχετικοί περιορισμοί για προϊόντα εταιρεών έξω από την Ευρώπη. Δεύτερο, το γεγονό ότι περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση, το brokering. Είναι σωστό να μην ασχοληθούμε μοναχά με την άμεση εμπορία, αλλά και με αυτού που κάνουν τους μεσίτε αυτές τι αγορα, αυτών των προϊόντων. Άλλη ερώτηση Μήπως πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο το πλαίσιο των προϊόντων που θα περιλάβει και βεβαίως και για τις χώρες που θα περιλάβει. Και θα υποβάλουμε και γραπτός προτάσεις, η μου δηλαδή, για την ενίσχυση του κανονισμού. Λούνες, ECR. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος υποστηρίζουμε, η ομάδα μου δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό τα όσα προτείνει η ίδια. Θεωρούμε κι εμείς ότι είναι θετικό που θέλει να διευκολύνει και να απλουστεύσει τις εξαγωγές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με ενισχυμένο έλεγχο των τελικών χρηστών και των τελικών χρήσεων. Λέγεται επίσης ότι τα μέτρα πρέπει να είναι όρθα σταθμισμένα. Για παράδειγμα, τα φάρμακα να μην περιορίζονται ακόμα και αν υπάρχει κίνδυνος καταχρησής τους. Το θηικό πεντονάτριο, για παράδειγμα, όπως λέει ένας ε, συνάδελφός μου που με επισήμανε, δηλαδή, επιλαμβάνεται σε ένα παράρτημα, και το οποίο χρησιμοποιείται ε, ως ε, πρώτο στάδιο της νάρκωσης, αυτό ε, πρέπει να μας αποσχολήσει. Μπορούμε να καλύψουμε τις περιπτώσεις αυτές που μας ενδιαφέρουν. Ίσως όμως να είναι απαραίτητο να εξετάσουμε ολόκληρο τον κατάλογο να δούμε ποια από τα φάρμακα αυτά που χρησιμοποιούν και σε άλλες χρήσεις. Πάντως, καταρχήν αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνεργασία με όλες και όλους τους συναδέλφους και βέβαια στο σχέδιο της Κομισιόν. Φορέντζα, Ενωτική Αριστερά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ, όπως και η συγγήτρια και οι προλήσαντες συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει καθόλου δευτερεύουσα σημασία. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωταγωνιστικό ρόλο για την αντιμετώπιση των βασανιστήριων και τη θανατική ποινή βεβαίω. Εμεί θεωρούμε ότι η καταπολέμηση των βασανιστήριων και άλλων ταπεινωτικών και απάθρων μεταχειρήσεων αποτελούν μια προτεραιότητα στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στι εμπορικέ και εξωτερικέ πολιτικέ. και οι χώρε μέλη πραγματικά έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να εξαλειφθεί το φαινόμενο του βασανιστήριων σε τρίτες χώρες. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο διμερείς ε, προσεγγίσεις και συμφωνίες, αλλά και πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε την ύπαρξη συγκεκριμένων απαντήσεων και προληπτικών για τα άτομα τα οποία υπόκειται σε βασανιστήρια. Σήμερα το φαινόμενο βασανιστήριων συνεχίζει να μεγεθύνεται εντός και εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν 134 επιχειρήσεις από την Κίνα που εμπλέκονται στο εμπόριο οργάνων που αφορούν αυτό το φαινόμενο και θα πρέπει να απαγορευτούν. 28 πριν κάποια χρόνια υπερτετραπλασιάστηκαν λοιπόν. Είναι μεγάλο επιχειρηματικό φαινόμενο τα βασανιστήρια. Περιλαμβάνει και στοιχεία κατά των ταραχών και για την τήρηση της δημοσίας τάξης. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να περιληφθεί δηλαδή στη σκέψη μας και να τον αντιμετωπίσουμε στις χώρες μέλη. Η επιχείρηση Sing Sing ε, εξήγαγε αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων ήδη και περιλαμβάνονται εδώ ήδη τα οποία επιφέρουν ηλεκτροσόκ σε διάφορα σημεία του σώματος, ευαίσθητα, γενικά όργανα κτλ. Γι' αυτό σε αυτά που θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να ενισχύουν τον κανονισμό του 2032 του 5, τον κανονισμό του Συμβουλίου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δούμε και το εμπόριο άλλου εξοπλισμού που αφορά την ασφάλεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εύκολα στα βασανιστήρια και σε αυτού του είδους συμπεριφορές. Ας πούμε τα όπλα τα οποία προκαλούν ηλεκτροσόκ σε άμεση ε, επαφή με το θύμα και άλλα που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην Αφρική και παράγονται στην Κίνα. Θα πρέπει να περιληφθούν εδώ στο κατάλογο των απαραγωμένων ειδών του κανονισμού. Επίσης, η διεθνής μεσολάβηση, ιδιαίτερα από Ευρωπαίους για αυτά τα είδη, ε, αποτελεί ένα σωστό μέτρο. Θεωρούμε όμως ότι είναι απαραίτητο να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά την ανάγκη απαγόρευσης δραστηριοτήτων προώθηση και διαθέσεων εμπόριου αυτών των αγαθών μέσω και της απαγόρευσης αυτών των ειδών σε όλες τις εκθέσεις και την πωλησή τους στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Θα πρέπει επίσης να ισχυθεί ο ίδιος ο μέσω της θέσπισης μιας συνολικής ρήτρα, ρήτρα catch all, ώστε να περιληφθούν, να επιτραπεί μάλλον σε όλες τις χώρες μέλη να να απαγορεύσουν μάλλον το εμπόριο ειδών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αλλά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα βασανιστήρια ή όπου υπάρχουν τέλο πάντων βάσιμε υπόνοιε ότι αυτά τα είδη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτού του σκοπού. Τέλο, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει πολυμερό την υιοθέτηση ενό αντίστοιχου κανονισμού για τον έλεγχο των ειδών εμπορικών ειδών βασανιστήριων διεθνώ. Και αυτό θα πρέπει να είναι από του κύριου πυλώνε τη πολιτική ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλε, η συναδελφό μου, βρίσκεται στη γερμανική Bundestag σήμερα, άρα κολλείται να είναι εδώ και γι' αυτό δεν μπορώ να προβώ σε σχόλιο. Begin, η FTD. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υπόγραψε λοιπόν διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες για την ε, κατάρριξη των βασανιστήριων στο εσωτερικό τους και επειδή είναι η πρώτη εμπορική δύναμη θα πρέπει να διασφαλίσει το ότι τα αγαθά που εξάγει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει εργαλεία για αυτό το σκοπό. Νομίζω όμως είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύεται με Πολλέ μη ευρωπαϊκέ χώρε που έχουν ήδη καταργήσει την θετική ποινή και τα ε, βασανιστήρια. Όμω πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι με τη σειρά του δεν θα επαναεξάγουν τα ίδια αυτά οι χώρε αυτέ, προς τρίτε χώρε. Και η τωρινή πρόταση τη Κομισιόν αφορά και του brokers, του Ευρωπαίου και όλου αυτού που παρέχουν ε, υπηρεσίε μεσολάβηση για αυτά τα προϊόντα, των οποίων η εξαγωγή και η εισαγωγή βεβαίω απαγορεύεται, επειδή αυτά τα ε, ήδη χρησιμοποιούνται μόνο για βασανιστήρια και θανατικές ποινές. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τα θέματα που αφορούν και τους εμπορευόμενους που μεταφέρουν αυτά τα είδη στην επικράτεια της Ένωσης χωρίς να έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες για τον τελικό τους σκοπό, τελική τους χρήση. Αυτό αφορά βεβαίω και τα τελωνία, αλλά και τις έχουμε κυρώσει στους εμπορικούς φορείς οι οποίοι παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες. Συμφωνούμε με την πρόταση, αλλά εμείς θα θέλαμε να τη βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μάργκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη παρουσίαση των βασικών θεμάτων που προκύπτουν από την πρότασή μας. Όπως είπε και η συγγήτρια, η πρόταση της Κομισιόν είναι να τροποποιήσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο εμπορικό κανονισμό του 2005 είναι ο 1236 του 5 για εμπορία συγκεκριμένων αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούν για θανατική ποινή, βασανιστήρια κτλ. Είναι τμήμα της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σχετίζεται και με την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες και είναι ο μοναδικός εμπορικός κανονισμός που περιορίζει το εμπόριο με μοναδικό στόχο να μην επιτρέψει τα ευρωπαϊκά αγαθά να χρησιμοποιηθούν για πραβιάς ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλα διεθνή εργαλεία απαγορεύουν και την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια χωρίς παρεκκλήσεις. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την θανατική ποινή είναι εξίσου απερίφραστη. Η θανατική ποινή καταργείται για όλα τα αδικήματα και είναι απαράδεκτη υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτές λοιπόν οι απόλυτες απαγορεύσεις ελήφθησαν υπόψη και ο 1236 του ρυθμίζει το εμπόριό μας με τις τρίτες χώρες. Απαγορεύει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές κάποιων αγαθών που βρίσκονται στον κατάλογο, όπως για παράδειγμα αγχώνες. Βέβαια υπάρχουν αγαθά τα οποία έχουν πολλαπλές χρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια άλλα αγαθά στον κατάλογο που υπόκεινται σε απέτηση εξαγωγικής άδειας έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να ελέγξουν την χρήση που θα γίνει αυτών των αγαθών από τρίτες χώρες. Ο κατάλογος ο ελεγχόμενος είναι τα μη θανατηφόρα όπλα, για παράδειγμα τα τέιζερ που προκαλούν ηλεκτρικό, ηλεκτροσόκ. Από το 2011 οι εξαγωγές και κάποιων φαρμακευτικών προϊόντων ελέγχονται, για παράδειγμα ανησυντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για εκτελέσεις μέσω θανατηφόρων ενέσεων. Η πρόταση της Κομισιόν για τροποποίηση του κανονισμού από τον Ιανουάριο πέρσι συμπεριλαμβάνει δύο νομικές πράξεις που προέκυψαν από μια αναθεώρηση που έκαναμε το 2011, με το 2012 και 2013. Η δεύτερη νομική πράξη είναι ο εφαρμοστικός κανονισμός 775 του 2014 που εκδόθηκε τον Ιούλιο και τροποποιεί τον κατάλογο των απαγορευμένων και ελεγχόμενων ουσιών. Εμείς αναθεωρήσαμε τα παραρτήματα 2 και 3 του 1236 του 5. Η πρόταση λοιπόν ε, αυτού του κανονισμού εστιάζει ε, στα προϊόντα τα φαρμακευτικά που βρίσκονται στον κατάλογο των ελεγχομένων προϊόντων και Κάναμε αυτές τις προσθήκες λόγω ετοιμάτων που λάβαμε από τα κράτη-μέλη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την κοινωνία των πολιτών. Μια χρονική στιγμή όπου ακούστηκαν πολλές ανησυχίες για το ότι φάρμακα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν για εκτελέσεις της ΕΠΑ. Όλα, κράτη, όλα τα κράτη-μέλη έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Και όπως είπα, η δική μας εξωτερική πολιτική δεν δέχεται την θανατική ποινή υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και αυτή είναι η διάκριση που κάνει, ε, που είναι μάλλον η διαφορά που μας διακρίνει από την ΙΠΑ για παράδειγμα και από την Κίνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καλύψουμε αυτή την νομοθετική πτυχή μέσω των δικών μας ε, κανονισμών. Με τον κανονισμό αυτό θέλουμε να είναι και καλύτερα εστιασμένοι οι έλεγχοι, ε, σύμφωνα και με τα όσα είπαν αρχικά σήμερα κάποιοι ευρωβουλευτές. Μια γενική απαγόρευση, για παράδειγμα, θα διευκολύνει το εμπόριο ε, με χώρες όπως είπα που δεν έχουν απαγορεύσει τη θανατική ποινή εδώ αναφέρομαι στο πρωτόκολλο 13 της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τροποποιήσουμε τους μηχανισμούς των ελέγχων ε, που ισχύουν σήμερα, δημιουργώντας δύο διαφορετικά συστήματα εξαγωγικών ελέγχων έτσι ώστε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούν για ε, εκτελέσεις, δηλαδή θανατική ποινή και για τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια. Ο κανονισμός του 5 δεν έκανε αυτή τη διάκριση και ο κατάλογος των ελεγχόμενων ουσιών τότε συμπεριλάβει μόνο τα αγαθά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια. Αυτή η κατανομή σε δύο συστήματα είναι απαραίτητη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρειάζεται σαφήνεια για, την, τον έλεγχο τελικής χρήσης που θα πρέπει να γίνει πριν χορηγηθεί μια εξαγωγική άδεια και δεύτερον για να λάβει υπόψη πως πολλές αλλά όχι όλες οι χώρες κατηρήσαν τη θανατική ποινή. Η τροπολογία στο μηχανισμό των εξαγωγικών ελέγχων δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξαγωγές κάποιων φαρμάκων, αλλά όλων των ελεγχόμενων αγαθών. Προτείνουμε πιο συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα, να επιτρέπουμε τη χρήση ε, μιας γενικής άδειας, όπως ε, χρησιμοποιείται στους εξαγωγικούς ε, ελέγχους για τα αγαθά διτής χρήσης και δεύτερον το πεδίο εφαρμογή των ελέγχων να διευρυνθεί για να καλύψουμε και την τεχνική βοήθεια και τις υπηρεσίες δια ε, μεσολάβησης όπως είπε και ο συνάδελφός σας. Θα πρέπει να μην επιτρέπεται η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών όταν ο προμηθευτής αυτής της υπηρεσίας έχει υπόνοιες ή γνώση πως τα σχετικά αγαθά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή ή για βασανιστήρια. Έχουν γίνει συζητήσεις στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και φάνηκε πως τα κράτη-μέλη Εν τω μεταξύ έδειξε μια προτίμηση για ένα σύστημα ε, εκ των προτέρων αδειοδότησης που θα είναι παρόμοιο με αυτό των εξαγωγικών ελέγχων. Η απάντησή μας ήταν πως για μας το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση και αν αυτό το πετύχουμε τότε θα μπορούσαμε θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δεχτούμε αυτή την προσέγγιση των κρατών μελών. Έχουμε ακόμα ένα θεσμικό θέμα που πρέπει να αναφέρω. Η πρόταση αυτή τη στιγμή ε, σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση αρμοδιότητες αποτελεί νεκρό γράμμα. Γιατί έχουμε πια τον κανονισμό 37 του 2014. Κάτι το οποίο συμπεριλάβαμε. Περάσατε το χρόνο σας. Μήπως μπορείτε να κλείσετε. Τελειώνω. Η επίγουσα διαδικασία είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα θέλαμε να διατηρηθεί γιατί θα μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε ταχύτατα την νομοθεσία σε νέα προϊόντα, για παράδειγμα, που κυκλοφορούν στην αγορά, φάρμακα, ε, τα οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε κτλ. Κλείνω λέγοντας, κυρία Πρόεδρε, πως όπως είδατε κι εσείς, είναι μία ε, πρόταση για την οποία υπάρχει μεγάλη προσμονή. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα ακολουθήσουμε τις ε, ε, προσπάθειες που κάνει η, Λιθουανική, με η Λετωνική Προεδρία για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Είχαμε επαφές μεταξύ της κυρίας Χάκια και της ε, Λετωνικής Προεδρίας. Είμαστε στη διάθεσή σας και θα διευκρινίσουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο εσείς θα μας ζητήσετε πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάκ έχει το λόγο για παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Να πω πως χαίρομαι που υπάρχει αυτή η κοινή μας δέσμευση για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Μία κοινή φιλοδοξία που καλύπτει όλα τα ε, θέματα αυτά, γιατί διαβάζουμε πραγματικά ανατριχές δικαιαστικές λεπτομέρειες για το πώς γίνονται τα βασανιστήρια στην πράξη. Πολύ σωστό είναι εδώ λοιπόν να αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και με οποιονδήποτε κανονισμό είναι σημαντικό οι πρακτικές που θα ακολουθήσουμε να μην ε, δυσκολέψουν όσους ε, χρειάζεται να εφαρμόσουν τους κανόνες μας και για τους γιατρούς και για τον ιατρικό κλάδο θα κάνω κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσω πως οι νόμιμες χρήσεις κάποιων ε, φαρμάκων, για παράδειγμα ε, κάποιων αναισθητικών, να μην ε, πληγούν από αυτή την νομοθεσία. Θέλουμε να αποφύγουμε μόνο την κατάχρηση ή την παραβίαση των όρων χρήσης αυτών των φαρμάκων όταν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα γενέσεις. Τώρα, κανονισμός ε, για τα βασανιστήρια, αν θα κάνουμε τη διάκριση αγαθάδη της χρήσης και κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια σας πληροφορώ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις σωστές επιλογές και έχω μια πρόταση ε, γραπτή την οποία θα σας μοιράσω. Ξέρω πως η ψηφοφορία είναι για τον Ιούνιο. Οπότε ελπίζω πως θα έχουμε κλείσει το θέμα πριν το τέλος της Προεδρίας και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με όσους επιθυμούν ε, να με βοηθήσουν στην ενημέρωση αυτού του κανονισμού. Προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο. 20 λεπτά μόνο για το επόμενο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει μια, εγκρίνει μια ανακοίνωση για τη στρατηγική για την προστασία της διανοητικής ε, ιδιοκτησία στις τρίτες χώρες. Το 2004 είχε η, με συγχωρείτε, είχε εγκριθεί το 2004, η νέα στρατηγική έχει μια διεθνή προσέγγιση, εξετάζει τις εξελίξεις, προτείνει λύσεις για να βελτιώσουμε τη δράση μας, για να προωθήσουμε πιο αυστηρούς κανόνες για θέματα διανετικής ιδιοκτησίας στο εξωτερικό και για να μην έχουμε εμπορία παραχαραγμένων αγαθών. 200 δις ευρώ χάνονται το χρόνο, υπολόγισε ο ΠΟΕ. Και στη στρατηγική αυτή ε, προτείνονται κάποια μέτρα για το 2015. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει στη συζήτηση. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Η κυρία Μόσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως σωστά λέγατε, ξεκινάμε σήμερα τη συζήτηση για την έκθεση πρωτοβουλία για την στρατηγική βάση τη στρατηγικής που παρουσίασε η Κομισιόν την 1η Ιουλίου του 2014 για την προστασία και επιβολή δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία μετά από την απόρριψη εκ μέρους του Κοινοβουλίου το 2012 της ΑΚΤΑ. Και σε γενικέ γραμμές θεωρούμε ότι το γεγονός ότι η Κομισιόν επαναπαρουσίασε και θέλησε να συνεχίσει την προσπάθεια προσδιορισμού της στρατηγικής της και της ενίσχυσης των δικαιωμάτων δικαιωτικής ιδιοκτησίας Θέλουμε ότι είναι πολύ θετικό και το συμμεριζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας αποφάσισαν να συντάξουν έκθεση τροπολογίας ακριβώς για να καταδείξουν τη σημασία που αποδίδουν όσον αφορά τον εντοπισμό της βέλτιστης στρατηγικής και πιο αποδοτικής. Μετά από μια τεχνική ενημέρωση και συναντήσεις με τους stakeholder που κάναμε πρόσφατα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι θεωρούμε σε γενικές γραμμές ότι η προσέγγιση της Κομισιόν είναι ισόρροπη και κυρίως υπογραμμίζουμε τη σημασία που δίδεται και ενισχύεται για τα δικαιώματα αυτά και την ίσχυσή τους στα πλαίσια των γενικότερων πολιτικών ενίσχυσης της οικονομίας μας και της οικονομίας τρίτων χωρών. Παρ' όλα αυτά παραμένουν κάποια στοιχεία με τα οποία διαφωνούμε, τα οποία θα προσπαθήσω να συνοψίσω στο λίγο χρόνο που έχω. Σε τρεις ομάδες θα αναφερθώ, χωρίς βεβαίως να είμαι διεξοδική για ένα τόσο ευρύ ζήτημα. Η πρώτη ομάδα παρατηρήσεων σε σχέση με τη στρατηγική της Κομισιόν αφορά την ανάγκη να κάνουμε όσο πιο συνεκτική γίνεται την προσέγγιση σε διάφορους τομείς. Καταρχάς δηλαδή η ανάγκη για συν... συνεκτικότητα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Και από αυτό γίνεται μεγάλη συζήτηση που αφορά την ενιαία αγορά και την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά και συνεκτικότητα μεταξύ πολιτικών που αφορούν το διεθνέ εμπόριο και άλλε πολιτικέ όπω οι πολιτικέ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, καταπολέμηση του ξεπλήματο, φοραποφυγή, απάτη κλπ. Τέλο, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα και συνοχή μεταξύ τη εμπλοκή όλων των stakeholder, ιδιαίτερα εκείνων που δεν είχαν την ίδια σημασία τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις καταναλωτών, για να αναφέρω μόνο κάποιες. Και η δεύτερη ομάδα παρατηρήσεων αφορά αντίθετα την ανάγκη στα πλαίσια στρατηγικής της Ένωσης προς τις τρίτες χώρες για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πολιτικών ώστε αυτές να είναι όσο πιο αποτελεσματικές γίνεται. Κατά την άποψή μας, στη στρατηγική δεν υπογραμμίζονται διόντως. Καταρχάς, όσον αφορά την γεωγραφική σκοπιά, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι καλύτερες πολιτικές για τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές που εξετάζουμε, γνωρίζοντας καλά ότι ο αντίκτυπος όσον αφορά την προστασία και την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων δεν είναι ταυτόσιμο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεύτερο σημείο. Η ανάγκη διαφοροποίησης μεγαλύτερης διαφοροποίηση μεταξύ φυσικών και ψηφιακών προϊόντων. Σημαντικό στοιχείο αυτό που θεωρούμε ότι θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε όσο πιο έντονα γίνεται. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό ακριβώς είναι ουσία του ζητήματος της στρατηγικής που συζητάμε. Και τρίτο σημείο, τρίτο σημείο που αφορά την ανάγκη διαφοροποίηση είναι η ανάγκη του να εντοπίσουμε τι προτεραιότητες που βρίσκονται στα γενικότερα πλαίσια των δικαιωμάτων ενωτική ιδιοκτησία, χρησιμοποιώντα όμω ταυτόχρονα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα που έχουμε στη θέση μα και το impact assessment, που μπορούν να αποβούν χρήσιμα όσον αφορά τον προσδιορισμό αυτών των προτεραιοτήτων. Τέλος, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι υπάρχει κάποια εντύπωση το ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις κάπως συστερούν δηλαδή δεν έχουν την ίδια με αυτοί που έχουν άλλα θέματα στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής. Σε εγγύησαμε πάντως όσον αφορά τη διαφοροποίηση μας λυπεί η έλλειψη μιας ε, διεξοδικής μελέτης για τους λόγους για τους οποίους απορριφθήκε η άκτα και για την ανάγκη βεβαίως να ξεκινήσουμε από εκεί ώστε να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη στρατηγική. Τελευταία ομάδα παρατηρήσεων αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτάθηκαν στη στρατηγική. Σε ελληνικέ γραμμέ συμφωνούμε με την προσέγγιση, Όμω δεν είναι σαφέ. οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να ευκαινιστεί περισσότερο, το με ποια νομιμότητα θα εφαρμοστούν σε αυτές οι συγκεκριμένε δράσεις σε σχέση με τρίτες χώρες. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από ένα moral dissuasion όσον αφορά την ε, υπογραφή διεθνών συνθήκων που ισχύουν, αλλά και εδώ χρειαζόμαστε έτσι περισσότερη ακρίβεια. Επίση είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε το πόσο η Κομισιόν θα δώσει τα κονδύλια και τους πόρου και ποιου πόρου θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν ώστε να κατανοήσουμε αν π.χ θα μπορούσαν να υπάρξουν ατασέ για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής Ιδιοκτησία σε διάφορες χώρες. Ή αντίθετα θα υπάρξει τέλο πάντων ένας συντονισμός ή χρήση των εκπροσώπων των χωρών εκεί όπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα άμεσα εκπροσώπηση τη Κομισιόν, help desk κτλ. Το πώ θα μπορούσε επίση να δώσει κανεί νομική αρρωγή όσον αφορά τι συμφωνίε με τρίτε χώρε κλπ. κλπ. Δύο τελευταία που νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω. Πρώτον, φάρμακα. Θεωρούμε ότι είναι θετική η προσέγγιση της Κομισιόν, δηλαδή να προχωρήσει στον κανονισμό, όμως σε αυτή την πρώτη φάση θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να δοθεί μέγιστη προσοχή στην ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των γενώσιμων και της αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας. Δεύτερο σημείο. Θεωρούμε θετικό το ότι δρούμε στα πλαίσια του ΠΟΕ για να ενισχύσουμε την στρατηγική προστασία δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας, όμως είναι σημαντικό εξίσου να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να περιληφθεί ένα κεφάλαιο σε όλους τους PR στις ημερείς συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε. Εδώ θα κλείσω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια θα ελέγξουμε περισσότερα χρήσιμα στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci, Monsieur Caspari, pour le PPE. Non. Euh, David Martin, non. τώρα κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Α, η κυρία Μακράρκιν θέλει να μιλήσει. Εγώ θα μιλήσω κυρία Πρόεδρε. Και πρώτα θα ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτές τις πρώτες σκέψεις που κατέθεσε για το σημαντικό αυτό το σχέδιο. Ένα από τους λόγους που θέλησα να γίνω μέλος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου είναι και αυτή η υπόθεση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας. Και μας πρέπει έχουμε την εργαλειοθήκη για να τα υποστηρίζουμε τα δικαιώματα αυτά όταν, όταν ε, προκύπτουν προβλήματα εκτός των συνόρων μας. Πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι υποστηρίζουμε τα ε, διανοητικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους καταναλωτές να πιστέψουν ότι είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό να κατεβάζουν από το διαδίκτυο ταινίες ή μουσική και ούτω καθεξής χωρίς να πληρώνουν τίποτε. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο με τα απαραίτητα μέτρα που να πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν αλλά και με εκπαίδευση του κοινού για το ότι πρέπει να πράττουν για να είναι καταναλωτές της σύγχρονης εποχής. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τρίτες χώρες. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική εκεί, αλλά και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, διότι δεν διαθέτουν την υποδομή ούτε τις ικανότητες για να επιβάλλουν σεβασμό της προστασίας των πραγματικών δικαιωμάτων στις επικρατείες τους. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να τις βοηθήσουμε για να βάλουν σε εφαρμογή τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να προστατεύσουν και τι δικέ του οικονομίε αλλά και τι δικέ μα βιομηχανίε. Και βεβαίω και η εκπαίδευση των ε, καταναλωτών αλλά και η συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, των stakeholder. Να συνεργαστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες μέλη για να κατανοήσουν τα προβλήματα, να ε, μοιραστούν τις πληροφορίες αυτές για τα προβλήματα που μπορούν και αναφύονται και ταχύτατα και αυτό είναι και το πρόβλημα. Είναι όλες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις που είναι θαυμάσεις μεν αλλά που δυστυχώς σημαίνουν ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν ταχύτατα και να μην μπορούμε να τα ε, εντοπίσουμε. Υπάρχει λοιπόν πρόταση της Επιτροπής στην οποία μπορούμε να βασιστούμε και εγώ ευχαρίστω θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια και με τις συναδέλφους μου εδώ αλλά χρειάζεται μια ευρύτερη αντίδραση και ένας ευρύτερος διάλογος. Πρέπει να θεσπιστεί μια στρατηγική οριζόντια. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Ενίας Αγοράς για να φτιάξουμε ένα σχέδιο δράσεως. Και βέβαια και με τους ε, βουλευτές μας που ασχολούνται με τα τελωνία. Εσείς κύριε Σόλτς. Η σκιώδη συγγήτριά μας, Αν Μαρή, με παρακάλεσε να παρουσιάσω τις απόψεις της για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Δεύτερη φορά τώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα προστασίας ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα είχαμε συζητήσει και για τους παρόχους ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Τώρα η συνάδελφος μου Ανμαρή τονίζει ότι το διαδίκτυο από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και με ταχύτατη ανάπτυξη όλο τον κόσμο οδήγησε και στην παγκοσμιοποίηση. Βεβαίως τεράστια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, όμως έχει ανοίξει και την πηξίδα της σε ό,τι αφορά το copyright. Δεν υπάρχει πλέον ε, καμία ε, διαφορά ανάμεσα στο πρωτότυπο και, στη, και στο αντίγραφο με, λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας. Τώρα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. Είτε με τον μεγάλο αδελφό, όπου παρακολουθεί όλα τα κομπιούτερ που μπαίνουν στο διαδίκτυο. Αυτό όμως σημαίνει περιορισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γραφειοκρατία, κόστος και θα προκαλέσει σημαντικότατες αντιστάσεις όπως δείχνουμε και με το νομοθέτημα Άκτα του 2012. Η Αν Μαρή λέει, εξετάζοντα την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτή τάσεται υπέρ μια άλλη προσέγγιση. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε αγοράζει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ένα άδειο CD, οτιδήποτε, πληρώνει ένα τέλος το οποίο πηγαίνει σε ένα κεντρικό ε, οργανισμό. Και από αυτά τα έσοδα του κεντρικού οργανισμού αποζημιώνονται μετά η παραγωγη Έτσι ενισχύουμε και το έργο του δημιουργού και βεβαίως διασφαλίζουμε ότι την αμοιβή τελικά ή την αποζημίωση θα την λάβει ο δημιουργός και όχι οι μεγάλες βιομηχανίες που διαμεσολαβούν. Αυτή η προσέγγιση είναι και πιο αποτελεσματική και πιο ε, δίκαιη και περιορίζει το λιγότερο δυνατόν την προσωπική μας ελευθερία. Αυτή είναι η πρόταση Σαν Μαρή και την καταθέτω. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Άλλος κανείς. Α, κύριε Πικίν. Σας ευχαριστώ. Η διαδοτική ιδιοκτησία αφορά την κοινοτομία και την ανάπτυξη. Τη χρειάζεται η Ένωση για να παραμείνει ανταγωνιστική με χώρε όπου το εργατικό κόστος είναι οπωσδήποτε χαμηλότερο. Οπότε στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα προωθήσουν την καινοτομία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μας δείξουν τον δρόμο εξόδου από την κρίση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η βιομηχανία της γνώσης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική Ευρώπη 2020. 8 δις απώλειες στο ΑΕΠ υπολογίζει ότι είναι η Ένωση της απομεμήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς σύγχρονο και ολοκληρωμένο που να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των χρηστών και των δημιουργών. Θεωρούμε απαραίτητο ότι τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να περιληφθούν στις συνθήκες υποδιαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μπορέσουμε να διακρίνουμε μεταξύ της προστασίας, πατέντες κλπ και των προνομίων που γίνονται μετά αποκλειστικά που φύγουν τον πολιτισμό, την υγεία ή την ελευθερία των ιδεών. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε υπερβολικοί με την προστασία των δημιουργών γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν παράτεπα από κάποιους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια προσέγγιση όχι ιδεολογική αλλά πρακτική και θα χαρώ να συνεισφέρω ως σκιώδης. Ευχαριστώ κύριος Γιασένη Κομισιόν. Πρώτα ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δύο βασικά σημεία. Τα σχόλια της εισηγήτριας για την διαφοροποίηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την διαφοροποίηση νομίζω είναι σημαντικό να διακρίνουμε και να διαχωρίσουμε αυτό το έγγραφο από το έγγραφο που υιοθέτησε η Κομισιόν που αφορά την εσωτερική πλευρά της εξίσωσης για την προστασία και επιβολή. Υπάρχει μια διτή σταδιακή εσωτερική και εξωτερική. Εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με την εσωτερική κυρίως. Και αυτό με οδηγεί στο σημείο που έθεσε ο κύριος ε, Σόλτς, συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί εδώ δεν θέλουμε να καταλάβουμε ή να λάβουμε θέσεις προκατηλημένες για αυτά τα ζητήματα. Δουλεύουμε βάσει της ισχύουσας και μελλοντική ευρωπαϊκής δημοθεσίας. Υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις που δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα θέματα και που δεν σχετίζονται με την ανακοίνωση που αναφέραμε γιατί έχουν να κάνουν με την εξωτερική διάσταση. Ένα δεύτερο σημείο για τον καθορισμό προτεραιοτήτων συμφωνώ γιατί δεν έχουμε ανεξάντηλους πόρους. Κάθε δύο χρόνια έχουμε μια έρευνα IPR που ολοκληρώνεται και θα ολοκληρωθεί και φέτος και λαμβάνουμε τις συμβολές και τις απόψεις των εμπλεκομένων, των χωρομελών, των φορέων κτλ. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καταρτίζουμε ένα κατάλογο και εντοπίζουμε τις κυρίες χώρες όπου παρουσιάζουν προβλήματα. Αλλά εμείς δεν έχουμε επαρκείς πόρους ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις χώρες του κόσμου. Και το πρώτο τρίμηνο θα έχουμε την νέα αυτή ανακοίνωση που θα καταρτήσει ένα κατάλογο προτεραιότητας για τα επόμενα δύο χρόνια και θα ενημερώνεται. Εδώ θα σταματήσω πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Μόσκα, εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ και στους αδέλφους, αλλά και την Κομισιόν για τις παρατηρήσεις. Μπορούμε να συνοψίσουμε λέγοντας ότι συμμεριζόμαστε το γεγονός ότι ξεκινάμε από κάποια θετικά στοιχεία που περιέχονται στην στρατηγική της Κομισιόν. Όλοι οι συνάδελφοι συμφωνούν σε αυτό και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της μελλοντικής μας δουλειάς. Να υπογραμμίσω μόνο δύο σημεία που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Αφενός, όπως είπα, κατά την πρώτη παρουσίαση το γεγονό ότι το πιο λεπτό σημείο θα είναι το να βρούμε μια σωστή ισορροπία για να προστατεύσουμε αφενός τους δημιουργούς και τους καταναλωτές των ψηφιακών προϊόντων αφετέρου. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που θα είναι το πιο δύσκολο να νομοθετήσουμε, ώστε να προστατεύσουμε όλους τους εμπλεκόμενους. Και αφετέρου και σε σχέση με αυτό το σημείο, αυτό που μόλις μας είπε, για αυτό που μόλις μας είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι αλήθεια ότι εμείς σήμερα μιλάμε για την στρατηγική που αφορά τρίτες χώρες και είναι αλήθεια ότι έχουμε την ευαισθησία να μην προκαταβάλουμε μελλοντικές αποφάσεις για την εσωτερική την ενιαία αγορά. Όμως δεν μπορούμε να μην θεωρήσουμε ότι αυτές οι δύο στρατηγικές δεν θα πρέπει να συμβαδίζουν και να μην θεωρούνται ένα ενιαίο πράγμα. Οπότε πολύ καλά να μην προκαταβάλουμε μελλοντικές αποφάσεις εσωτερικές, όμως για να είναι αποτελεσματικές στρατηγικές εμείς θα πρέπει τις δύο συζητήσεις αυτές να τις κάνουμε εκ παραλέλου. Όλοι μας νομίζω θα συμμετάσχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Για το χρονοδιάγραμμα, η επόμενη εξέταση της έκθεσης θα γίνει στις 18-19 Μαρτίου, στην επόμενη συνέντευξη της Επιτροπής μας, 23 Μαρτίου στις 5 ώρα το απόγευμα κατάσταση τροπολογιών, με ψηφοφορία Απρίλη ή Μάη και στην Ολομέλεια στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο σημείο στην ημερησιά μας. Ευχαριστώ τους διερμηνείς που μας παρέχουν πέντε λεπτά παραπάνω. Θα είμαι πολύ γρήγορη. Δεστηριότητε της ομάδας παρακολούθησης. Τίζα, κυρία Ρέντινγκ, η ομάδα παρακολούθησης σύλθε σήμερα πριν τη συνεδρίασή μας για τον 11ο κύκλο διαπραγματεύσεων ΤΙΖΑ και συγκεκριμένα για τρεις τομείς προβλέπετε μια δημόσια κρόση για το τι αύριο το πρωί. Έχετε να πείτε κάτι κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Όπως είπατε σωστά. Είχαμε την τρίτη συνάντηση τη ομάδα παραγωγής μόλι σήμερα. Συνάντηση όπου είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τους κύριους διαπραγματευτές, με τον κύριο διαπραγματευτή. Μας είπε ότι αυτό που συζητήθηκε είναι το αποτέλεσμα του 7ου γύρου διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Η Ουρουγουάη συμμετέχει τώρα στις διαπραγματεύσεις, οπότε είμαστε 24. 24 μέρη. Στην Τίζα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως ένα. Συζητήσαμε μία που αφορούν τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν την, προτιμούμενη, πιο προτιμούμενη χώρα και το θέμα της πρόσβασης στις αγορές που δεν θα ρυθμιστεί άμεσα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να θέσουμε ένα, μια σαφή περίμετρο για τις διαπραγματεύσει. Και υπάρχει η βούληση για να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κλπ. Ο επόμενος γύρος θα είναι τον Απρίλιο, ώστε να προχωρήσουμε με τρόπο πιο δομημένο. Μας ενημέρωσαν ότι η αποτίμηση θα γίνει φέτος ώστε να επιταχυθούν οι συνομιλίες και πρόεδρε τότε ακριβώς θα είναι η στιγμή όπου και εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της διαδικασίας στην Επιτροπή μας. Στη σημερινή συνεδρίαση οι εκπρόσωποι της Κομισιόν μας έδωσαν πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς δεδομένων, υπηρεσίε, χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε κτλ. Προέλευση χωρική των δεδομένων συζητήθηκε με τρόπο επικοδομητικό στα πλαίσια τη ημερησία διαταξή μα. Συζητήσαμε επίση το θέμα τη πρόσβαση σε τηλεπικοινωνικέ δομέ σε τρίτες χώρες και την ανάγκη να μην υπάρχουν διακρίσεις από τις διατάξεις στην Ένωση. Μιλήσαμε επίσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την πρόσβαση στις αγορές και σχέση με διεθνείς προδιαγραφές όπως η Βασιλεία 3. Πρόεδρε, είπατε ότι αύριο το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε βάθος περισσότερο για αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης για την ΤΙΖΑ. Ευχαριστώ. Βιετνάμ τώρα. 29 Γενάρη συνεδρίαση ομάδα παρακολούθηση ο κ. Ζαρανίου, ο ναι, όντω πρόεδρε. Στις 29 του Γενάρη συνεδριάσαμε. επόμενο γύρος διαπραγματεύσεων για το συγκεκριμένο θέμα το Μάρτι εντάξει 9 και 19 κάπου και προετοιμάζουμε και τη συνάντηση με το Βιετνάμ στι αρχές του Απρίλη. Είχαμε, θα έχουμε τον πρεσβευτή τους, συν το κύριο διαπραγματευτεί. Αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε και έτσι, κάποια έτσι καυτά ζητήματα που αφορούν εκείνε τι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ομάδα Καναδά, ΙΠΑ, Ρωσία, Νότιος Κορέα, Μεξικό και Μαγκρέπ Επίση συνεδρίασαν. Αυτά συνάδελφοι, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνει η συνεδρίαση για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Σα ευχαριστώ. Γεια σας.